even Μ' αρέσει που σας βλέπω να τσομπολεύετε μεταξύ σας, αλλά μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Καλώς ήρθατε μετά από τις ψηφοφορίες και καλώς ήρθαν και οι αναφέροντες κυρίως. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο θα δείτε και οι διερμηνείς θα διαβάσουν κάνοντας αυτόματη μετάφραση χωρίς να ακούνε την, ε, τον ήχο. Δεν βοηθάει. Το κάνουμε αυτό επειδή σεβόμαστε τον κόπο στον οποίο μπήκαν τα ξέδους μέχρι εδώ οι αναφέροντες. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την 2563 αναφορά σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Ισπανίας. Έχουμε την, και τα στεγαστικά. Έχουμε τον Χωσέ Λακάλ Μάρκες από την Ισπανία. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Καλημέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών που μας ε, έκανε δεκτό το αίτημα για τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα λύσει με δεσμευτικό τρόπο τις καταγγελίες και τις προσφυγές των πολιτών κατά των τραπεζικών καταχρήσεων. Πάνω από 40.000 πολίτες στήριξαν το αίτημα αυτό με συλλογή υπογραφών στο change.org. Τρεις είναι οι στόχοι στην αναφορά μας, να βελτιώσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, να είναι πιο δίκαιο δηλαδή και διαφανές, να προασπίσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και να αποφύγουμε την κατάρρευση των δικαστηρίων. Τον Απρίλιο 2015 ζητήσαμε από το να πάψουν να ισχύουν οι ρήτρε καθορισμού ενός ορίου στα ε, επιτόκια των στεγαστικών δανείων και την επιστροφή των ε, αχρηστούς καταβληθέντων ποσών και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επίπεδη μετά από το Β80755 2015 επειδή δεν ήταν από τα μέτρα αποτελεσματικά να παρακολουθεί την ε, εφαρμογή των νέων μέτρων. Έχουμε ένα, διάγραμμα, ένα βασιλικό διάταγμα τον Ιανουάριο 2017 για επίγοντα μέτρα προστασία των καταναλωτών και εκεί αποφασίστηκε ότι αν ε, υπάρχουν ε, τέτοια χρωστή καταβληθέντα ποσά θα πρέπει οι τράπεζε να αποφασίσουν αν θα τα δώσουν πίσω ή όχι και έτσι κάθε τράπεζα έκανε ό,τι ήθελε, ιδίω όταν αποφάσιζαν να επιστρέψουν χρήματα δεν έδιναν το σωστό ποσό γιατί το διάταγμα δεν είναι ξεκάθαρος προς ε, το ντόκο υπερημερίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται. Εμείς ε, έχουμε στραφεί σε πραγματογνώμονες και κάνουμε μελέτες και όποτε βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια ενημερώνουμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Τράπεζα της Ισπανίας. Και μας λένε ότι θα μπορούσε να επιβληθεί στο Foundation U-Bank ε, πιθανό πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι παράδοξη η τράπεζα ε, της Ισπανίας να μπορεί να ε, επιβάλλει πρόστιμα σε ένα ίδρυμα που θέλει να προασπίσει τους πολίτες από τις καταχρήσεις των τραπεζών αλλά δεν μπορεί να τιμωρήσει καμία τράπεζα για την καταχρηστική αυτή πρακτική. υπάρχουν από ό,τι φαίνεται πάνω από 200.000 δικαστικά αιτήματα τα οποία έχουν κατατεθεί λόγω αυτών των επιτοκίων και υπάρχουν και 17.000 αποφάσεις υπέρ των πολιτών κατά το 97% των περιπτώσεων. Πέρα όμως από αυτή τη ρήτρα έχουμε βρει πάνω από 30 καταχρηστικές ε, τέτοιες ρήτρε και κακές τραπεζικές ε, πρακτικές που εξακολουθούν να εφαρμόζονται εν γνώση της Τράπεζας Ισπανίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί όμως καμία κύρωση και δεν έχει ληφθεί κανένα πρόστιμο στους παραβάτες, ούτε έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για να διορθωθούν. Πέρα λοιπόν από αυτή τη ρήτρα έχουμε ότι όλα τα έξοδα τα ε, αναλαμβάνουν οι πελάτες, δηλαδή αμοιβή για δέσμευση κεφαλαίου μελέτης, για αναδοχή χρέους, ε, για την ε, πρόορια κύρωση, πληρωμή των φόρων, συμβολογραφικά έξοδα, έξοδα καταγραφή στο κτηματολόγιο, διαχείριση, εκτίμηση, στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Δεν μπορεί να επιλέξει ο πελάτης το σύστημα απόσβεσης του δανείου. Έχουμε την ρήτρε 365 κάθετος 360 ημέρες, έχουμε με πολλών, πολλαπλών νομισμάτων δάνεια. Έχουμε το δίκτυ IRPS, ε, την ε, τόκου υπερημερίας, επιβολή των εγγυητών, ε, ένσταση διζήσεως από τους εγγυητές δεν λαμβάνεται υπόψη. Ταχυδρομικά έξοδα, η προμήθεια για τη δανειακή χρωστική θέση, για τη λήξη, την εκ των λήξη, την ε, ρήτρα απαγόρευση άσκηση επαγγελματική δραστηριότητα στο ακίνητο. Ε, δεν υπάρχει δικαίωμα κοινοποίηση σε περίπτωση αναδοχής του χρέους, επιλογή δικαστηρίου κτλ. Επίσης, άλλες κακές πρακτικές τραπεζικές είναι ότι δεν υπάρχει νομιμοποίηση ό,τι αφορά ε, αυτές τις ε, πράξεις, καθότι πολλές φορές το ακίνητο δίνεται, μάλλον το δεν δίνεται σε ε, ταμεία επιθετικά αρπακτικά και επίσης δεν γίνεται σωστά η καθάριση των επιστροφών. Δεν θα πρέπει να λυθούν από τα δικαστήρια αυτά τα θέματα και γιατί είναι το κόστος μεγάλο για τον πολίτη, αλλά και γιατί υπάρχει καθυστέρηση στα δικαστήρια δικαστήρια και μπορεί να υπάρξει κατάρρευση του δικαστικού συστήματο. Ε, Επομένω, θεωρούμε ότι η δημόσια εξουσία είναι αυτή η οποία θα πρέπει με σαφεί νόμου ε, και αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου και εποπτεία να επιλύσει αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό λοιπόν και ζητούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να προβείτε σε μια πρόταση για τη δημιουργία οργανισμού, ο οποίο με δεσμευτικό τρόπο θα ε, λύσει το πρόβλημα και θα εξετάσει τι προσφυγέ των πολιτών κατά των ε, καταχρήσεων των τραπεζών και κάτι άλλο σημαντικό. Ε, μία διάσωση, θέλω να σα προτείνω, όχι οικονομική όμω. Διάσωση εντό αγωγικών τη εμπιστοσύνη των πολιτών που την έχουν χάσει πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Gracias a vuestro apoyo en la petición, tribunales exactly. y las instituciones europeas, la banca tiene que devolver los importes cobrados indebidamente por la aplicación de las cláusulas. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν πίσω ε, τα ε, κονδύλια, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες. Ε, πώς υπολογίζονται, ποιος πρέπει να τα επιστρέψει, ποιοι είναι αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν, θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή η πρόταση της τράπεζας. Ο μη πραγματικότητα είναι ότι κάθε τράπεζα στρέφει τα ποσά με δικά τη κριτήρια. Δεν υποχρεώνεται η τράπεζα να το κάνει σωστά και στι περισσότερες φορές τα ποσά που επιστρέφονται δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Ποια είναι τα λάθη των τραπεζών. Δεν επικαιροποιούν το κεφάλαιο που δεν πληρώνουν αποζημίωση ούτε εφαρμόζουν το τόκο υπερημερίας. Αυτό σημαίνει ε, και πάνω από το 50% του προσεπιστροφή επιστροφή πόσο γιατί δεν υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή η οποία με θεσμευτικό τρόπο θα ε, εξετάσει τις προσφυγές. Θα συνεχίσουμε τη δική σας βοήθεια να καταδικάζουμε τις ε, καταχρήσεις αυτές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάνω από 40.000 πολίτες στηρίζουν την αναφορά μας για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα που δεσμευτικά θα λύσει το πρόβλημα και θα ασχοληθεί με τις προσφυγές των καταναλωτών. That's a very informative video. Very good. I wish all the videos would be like... Πολύ ενδιαφέρον ε, βίντεο. Ελπίζω όλα τα βίντεο να ήταν έτσι, περιεκτικά, να τονίζουν ε, το ε, νόημα και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, Ρόμπερτ Ματιακ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τους διερμηνείς. Η αποζημίωση όλων των πληρωμένων ποσών είναι ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει πολλούς καταναλωτές και ίσως είναι και ορθό είναι πρόβλημα το γεγονός ότι δεν έχει επιληθεί ακόμα Κατά τη γνώμη μας δεν μπορούμε να σχολιάσουμε ακριβώς το, το τι ποσά είναι αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσουν οι τράπεζες, όμως είναι ξεκάθαρο ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση που έχουν πληρώσει παραπάνω ποσά ε, λόγω ε, λαθασμένων ε, ρητρών. Οπότε επίσης είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και το γεγονός ότι οι διαρθρωτικοί μηχανισμοί που έχουν εισαχθεί από την Λέω Κρέτο λέει από το 2017 έχουν οδηγήσει σε συμφωνίες μεταξύ καταναλωτών και τραπεζών και σε πάνω από 500.000 υποθέσεις που προαλείπτουν πάνω από 2,3 δις ευρώ και αυτές είναι δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες. Ταυτόχρονα ισχύει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει υπάρξει συμφωνία και οι τράπεζες έχουν αρνηθεί να επιστρέψουν τα ε, υπερβολικά πληρωμένα ποσά η βασική δυσκολία είναι ότι σύμφωνα με το δίκαιο της Ισπανίας οι συγκεκριμένες ρήτρες δεν είναι κατά ανάγκη άδικες. Αυτό συμβαίνει μονάχα σε περιπτώσεις που οι τράπεζες δεν ανταποκρίνονται σε ορισμένους κανόνες διαφάνειες. Και σε περιπτώσεις που οι τράπεζες έχουν αρνηθεί να επιστρέψουν τα αντίστοιχα ποσά, βασίζονται στο ότι ε, συμβαδίζουν ε, με, τις, με τους κανόνες διαφάνειες, το οποίο μπορεί βέβαια ε, να το αμφισβητήσουν οι καταναλωτές. Και βέβαια είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να το κρίνουν τα δικαστήρια σχετικά με το αν ισχύουν αυτές οι περιπτώσεις. Τώρα, η κυρώσεις ε, που προβλέπονται από την ε, οδηγία είναι ότι οι άδικοι κανόνες των συμβάσεων δεν είναι δεσμευτικές στις συμβάσεις αυτές, το έχει ξεκαθαρίσει το δικαστήριο και υπάρχει δικαίωμα αποσμίωσης. και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ε, τα, τα απαραίτητα ε, μέσα αποζημίωσης. Ο τρόπος ή αυτός σε περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν μπορούν να συμφωνήσουν ε, είναι η δικαστική οδός. Υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο όριο για τους καταναλωτές, όμως όσον αφορά το συμβατικό δίκαιο θεωρώ ότι η συνήθις διαδικασία είναι αυτή. Επίσης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας υπάρχει μια οδηγία ε, σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών και η οδηγία αυτή Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ε, τις ε, διαφωνίες τους ε, σε εναλλακτικά σώματα επίλυσης διαφορών και αυτό ισχύει και για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η Ισπανία από πλευράς της έχει ένα τέτοιο σώμα Όμως η οδηγία αφήνει στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν εάν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συμμετέχουν εθελοντικά ή υποχρεωτικά ε, σε τέτοιους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Οπότε η δημιουργία τέτοιων μηχανισμών όπως προτείνεται από την αναφορά είναι ίσως κάτι θετικό, ένα μέτρο το οποίο ίσως θα μπορούσε να επιλύσει περισσότερες υποθέσεις. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η οδηγία δεν, δεν απαιτεί κάτι τέτοιο. Ισχύει λοιπόν ότι αρκετές υποθέσεις βρίσκονται ακόμα ε, στα ισπανικά δικαστήρια. Αρκετές έχουν ε, κατατεθεί στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσης ε, και περιμένουμε περαιτέρω αποφάσεις τους επόμενους μήνες. Από πλευρά της Επιτροπής λοιπόν έτσι έχει η κατάσταση. Δεν παρατηρούμε επίσης το τι συμβαίνει ε, σχετικά με τις ε, ρήτρε και θα αντιστοιχώς θα ενημερώσουμε τις ε, Ισπανικές Αρχές. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστούμε πολύ και είναι πραγματικά ενδιαφέρον να μπορούμε να ακούμε και κάποιον που έχει μια φιλοσοφική προσέγγιση. Δεν μας συμβαίνει πολύ συχνά και όταν συμβαίνει είναι πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε τώρα να ακούσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Μπέτρις Μπεσέρα πρώτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του εκπροσώπου της μετά από αυτά που μας είπε ο κύριος Λακάγια από την Ισπανία και θέλω να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες ε, και να τους συγχαρώ που με πάρα πολύ αξιοπρέπεια και υπευθυνότητα συνεχίζουν τον αγώνα τους. Ε, έχουν κατατεθεί δεκάδες χιλιάδες ε, αιτήματα ακύρωσης της ρήτρα αυτής επιβολής ορίου στα και αυτό, αυτής καταχρηστικής ρήτρα που λέγεται κλαούς σουέλο στα ισπανικά. Τώρα έχουμε τις προτάσεις των τραπεζών τραπεζών που φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται στα ποσά που θα πρέπει να επιστραφούν κανονικά. Και υπάρχει αυτή η εγγύηση που προτείνεται, ο ειδικό οργανισμό δηλαδή, ώστε να είναι τα ποσά αυτά αναλογικά και να καταβάλλονται ω δι. Αυτό είναι το δίκαιο, διότι αυτέ οι καταχρήσει από πλευρά τραπεζών δεν είναι μόνο ισπανικό παράδειγμα. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να παρακολουθείτε ευρωπαϊκά το θέμα αυτό τη κατάχρηση τραπεζών. Αυτέ οι καταχρηστικέ τραπεζικέ πρακτικέ είναι ένα θέμα που πλήττει πολλέ χώρε. Ευχαριστώ και υπάρχουν ε, τα ε, διάφορα νομοθετήματα τα οποία επιβάλλουν στις τράπεζες να δράσουν διαφορετικά. Έχουμε ζητήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωση. Θέλουμε να υπάρξει επίσης καλύτερη εκπαίδευση για αυτά τα χρηματοοικονομικά θέματα. Είναι σημαντικό. Θέλω να υπενθυμίσω ότι και οι προσφυγές των πελατών, των τραπεζών φυσικά και δεν μπορούν να, να βρουν μια δεσμευτική λύση από πλευρά ε, τη Κομισιόν. Δεν υπάρχει μια κατεξοδότηση πράξη. θέλω να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και θέλω να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξετάσουμε ε, την, ε, τη ιδέα που προτείναμε. Μου φαίνεται καλή ιδέα τη δημιουργία του οργανισμού. Δεν ξέρω αν χρειάζεται όμω να γίνει μια μελέτη για να δούμε κατά πόσον αυτό μπορεί να γίνει και να λειτουργεί σωστά ένα τέτοιο οργανισμό. Μπορεί να υπάρξει κάποια εγγύηση ώστε οι συμπολίτε μα να έχουν ασφάλεια δικαίου Ιδίω όταν αυτό αφορά ε, την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους, τα οποία αναγνωρίζει ήδη η δικαιοσύνη. Και αυτά πρέπει να γίνουν σεβαστά στην πράξη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ Μπεατρίθ. Μαριά, ε, κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να συγχαρώ τους αναφέροντες διότι το θέμα που θέτουν παρότι επικεντρώνεται στην Ισπανία αφορά ουσιαστικά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε σε όλα τα κράτη. Αυτό που είδαμε ήταν ότι την ώρα που οι τράπεζες βρέθηκαν σε πρόβλημα κυρίως στην Ελλάδα, στην Ισπανία επίσης, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία τι έγινε έγινε μια μαζική δανειοδότηση οι πολίτες και τα κράτη έσωσαν τις τράπεζες και τώρα που οι τράπεζες έχουν σωθεί επιτίθενται κατά των καταναλωτών κατά των δανειοληπτών προκειμένου να εξοφλήσουν υποτίθεται οι δανειολήπτες τα χρέη τους. αυτό είναι κοινωνικά απαράδεκτο το οποίο συμβαίνει. δεύτερο ενώ υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί ένα μοντέλο ούτως ώστε όταν οι τράπεζες πωλούν τα δάνειά τους στα επιθετικά funds να μπορεί και ο δανειολήπτης να αγοράσει το δάνειό του στο ποσό που θα πωλήσει η τράπεζα το δάνειό του στα επιθετικά funds. Αυτό είναι το κυπριακό μοντέλο όπως λέγεται και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δίκαιο να μπορεί να συμβεί. Το τρίτο είναι να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να ιδρυθεί ένα ταμείο σωτηρίας δανειοληπτών με χρήματα τα οποία έχουν λάβει τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε αυτό το ταμείο να μπορεί να αγοράσει τα δάνεια των δανειοληπτών στην τιμή που πολλούνται στα επιθετικά φάντς και με αυτόν τον τρόπο να γίνει διευκόλυνση στους δανειολήπτες να σώζουν τα σπίτια τους. Το επόμενο θέμα το οποίο είναι αν θέλετε απαράδεκτο είναι ότι μια τράπεζα που έχει ένα ενυπόθηκο δάνειο βγάζει στον πληστηριασμό την πρώτη κατοικία, πουλάει το σπίτι, αλλά επειδή οι τιμέ των ακινήτων σε όλε τις ευρωπαϊκέ χώρε και στην Ελλάδα έχουν πέσει, σημαίνει ότι και ο δανειολήπτης χάνει το σπίτι του και μετά χρωστάει άλλα τόσα στην τράπεζα για να εξοφλήσει το δάνειο. Εγώ θεωρώ δίκαιο ότι από την ώρα που η τράπεζα πάρει το σπίτι του δανειολήπτη και το εκποιήσει με πληστηριασμό, να εξοφλείται και η απέτηση απέναντι στην τράπεζα. Άλλο θέμα που έθεσε ο αναφέρουν είναι το θέμα με τους εγγυητές. Οι εγγυητές πολλές φορές δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την ένσταση διζήσεως. Δηλαδή να πούνε στην τράπεζα να πάει πρώτα να εξοφληθεί από τον πρώτο φιλέτη και αν δεν εξοφληθεί τότε να ασκηθεί η αγωγή κατά του εγγυητή. Διότι ιδίω στην Ελλάδα έχουν βάλει τους εγγυητέ και παρετήθηκαν από το δικαίωμα διζήσεως. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για τους εγγυητέ. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί από ό,τι είδα την Ισπανία, αλλά απασχολεί πάρα πολύ την Ελλάδα και θα πρέπει και στο θέμα αυτό να υπάρχει μια παρέμβαση για να υπάρξει στήριξη των εγγυητών. Άλλο επίσης αντικοινωνικό θέμα είναι το εξή: Ενώ κάποιο έχει πάρει ένα δάνειο για ένα σπίτι το οποίο κατά 90% οφείλει στην τράπεζα έρχεται το κράτος και του απαιτεί να πληρώσει φόρο ακίνητης περιουσίας. Αυτό που στην Ελλάδα λέγεται ένφια. Και ενώ το σπίτι δεν είναι δικό σου, δεν είναι του δανειολήπτη, μια και η τράπεζα κατά 90% ε, το κατέχει έχοντας την υποθήκη, στο τέλος πληρώνει την, τον, φόρο ακίνητης περιουσίας ο δανειολήπτης χωρίς να δικό του το σπίτι. Αυτά λοιπόν όλα, μαζί με τις προτάσεις που έγιναν, πρέπει να τεθούν στο τραπέζι. Διότι εδώ γίνεται μια κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους των τραπεζών, έχουμε παραβιάσεις των δικαιωμάτων των καταναλωτών και εγώ βρίσκω καλή ιδέα αυτό που αναφέρθηκε, μια ανεξάρτητη αρχή, ίσως σε κάθε κράτος, ίσως πανευρωπαϊκά, να μπορεί να εξετάσει τα θέματα αυτά για να υπάρξει μια στήριξη των δανειοληπτών. Διότι οι δανειολήπτες έχουν αυτό το πρόβλημα και οι δανειολήπτες είναι στην μειονεκτική θέση. Επίσης δεν κάνει τίποτα ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε οι κεντρικές τράπεζες, είτε της Ισπανίας, είτε η Τράπεζα της Ελλάδος για την Ελλάδα. Αυτά λοιπόν τα σημαντικά θέματα πρέπει να τα δούμε, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, να εξετάσουμε την πρόταση των ε, δανειοληπτών και ίσως στο μέλλον να ετοιμάσουμε και εμείς μια δημόσια ακρόαση για την προστασία των δανειοληπτών, ιδίω όσων έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια πρώτη κατοικίας και εδώ η Επιτροπή μας να το δει το θέμα αυτό κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άχελα Βαλίνα. Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον αναφέροντα για την προσπάθεια, για την παρουσία που μας έκανε σήμερα και για τον αγώνα γενικά που δίνει μεταξύ άλλων βέβαια. Εμείς φυσικά ως Κοινοβούλιο πρέπει να μελετήσουμε την πρόταση των αναφέροντων και να δούμε τι μέτρα μπορούν να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο, γιατί πραγματικά είναι τραγική η εικόνα που δίνει η χώρα μου τουλάχιστον ε, στο εξωτερικό. Γιατί δεν προστατεύονται παρκώ τα δικαιώματα των καταναλωτών και γιατί φαίνεται να υπάρχει συνενοχή ε, των κυβερνήσεων ε, των εκάστοτε και ε, με τις τραπεζικές ε, ε, αρχές, με τις τράπεζες, δηλαδή που βλέπουμε να υπάρχει η απόφαση του δικαστηρίου που είναι θετική για τον δανειολήπη, για τον καταναλωτή και αμέσως συγκαλείται η ολομέλεια του ανώτατο δικαστηρίου και ακυρώνεται η απόφαση ουσιαστικά. Και τελικά την πληρώνει ο καταναλωτής. Εγώ πραγματικά λυπούμαι που οι Ισπανοί πολίτες συχνά πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια και ιδίως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να προασπιστούν τα δικαιώματά τους ε, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Έχουν υπάρξει πολλές νομοθετικές αλλαγές στην Ισπανία. Πάντοτε όμως ε, ε, μετά από κάποια απόφαση, αλλά χρειάζεται πλέον μια νομοθεσία που θα προστατεύει πραγματικά τους καταναλωτές σε όλους τους τομείς, σε όλες τις πτυχές και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα υπόθηκα Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, προφανέ αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να, μας να απαντήσει, μάλλον στου γραπτό, σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα μετά την ανάλυση τη ε, διαδικασία παραβάση ε, που έχει κινηθεί κατά τη ε, Ισπανία και επίση να σταλεί επιστολή στι Ισπανικέ Αρχέ για να ενημερώσουν σε σχέση με τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμόσει για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών αυτών πρακτικών. Ευχαριστώ, Μιράντα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίω προ τον αναφέροντα βέβαια που ήρθε εδώ. Δεν είναι δυστυχώ η πρώτη φορά που έρχονται αναφέροντε εδώ με τέτοια θέματα. Από το 2013 στην Επιτροπή μας ε, ε, βλέπουμε να έρχονται μέλη τη πλατφόρμα για τα ενυπόθηκα δάνεια ενό καταναλωτών ε, και έχουμε εξετάσει πολλές ε, υποθέσεις, πολύ αποκαλυπτικές για τις καταχρήσεις που γίνονται από τις ισπανικές τράπεζες και βλέπουμε και ότι σιωπούσε και η κυβέρνηση Ραχώη απέναντι σε όλα αυτά. Όταν ε, ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση, το δικαστήριο άρχισε να αποκαλύπτει ε, κάποιες τέτοιες πρακτικές, καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές. Η Ευρώπη ήταν αυτή η οποία έδωσε τη δυνατότητα ουσιαστικά στους καταναλωτές να απαιτήσουν ε, την, ε, το σεβασμό των δικαιωμάτων τους ε, που έφερε στο προσκήνιο το θέμα αυτό και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έτσι ξεκίνησαν και οι αλλαγές στην νομοθεσία ιδίως στην περίπτωση αυτή των καταχρηστικών αυτών ενυπόθηκων δανείων. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε στο πλευρό των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιστροφή ε, των ε, ποσών που κατέβαλαν ε, χρεωστήτως οι καταναλωτές στην τράπεζα είναι κάτι πολύ σωστό. Η ανάγκη αυτό να αποτελέσει προηγούμενο για τις μελλοντικέ περιπτώσεις όπως έγινε με την περίπτωση της Αμπάνκα στην Κορούνια που θέτει προηγούμενο η απόφαση του δικαστηρίου και σε πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου. Το θέμα είναι οι δανειολήπτες, 8 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι, δεν είναι λογικό να πρέπει αυτοί να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Για ένα τόσο βασικό ζήτημα, όπως είναι ε, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Δεν έχει επιληθεί υπόθεση. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις που αφορούν, αναρρύθμουν αριθμό δανειοληπτών και είναι και γιγαντιές οι οικονομικές επιπτώσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να καταγγείλουμε όλα αυτά που έγιναν. Με αυτό που είπε η κυρία Βαγίνα για το δικαστήριο και τον τρόπο που δρά. Και θα πούμε και το εξής. Ε, στην Ισπανία δεν προστατεύονται παρκώ οι καταναλωτέ. Μακάρι να αλλάξει αυτό. Όμω ε, είναι καταχρηστική, ε, κατ' εξακολούθηση η συμπεριφορά των τραπεζών. Υπάρχει ένα λόμπι ουσιαστικά που επηρεάζει και το βλέπουμε και στην περίπτωση των δικαστών με αυτά που έγιναν με τι αποφάσει σε κάποιε εβδομάδε τώρα ε, του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή αναφορά λοιπόν, ζητούμε να σταλεί επιστολή στι Ισπανικέ Αρχέ, αλλά και κάτι περισσότερο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε επάφη με το δικαστήριο από πλευρά Κοινοβουλίου δηλαδή ε, ώστε να ενημερώσουμε και να πούμε ότι δεν είναι μεμονωμένες αυτές ε, οι υποθέσεις. Πρόκειται για μια συνολική απάτη η οποία πλήττει πάνω από 8 εκατομμύρια καταναλωτές. Και από την άλλη πλευρά ζητούμε, όπως είχαμε ζητήσει και από το Διευθυντή τότε των χρηματοοικονομικών ε, θεμάτων και στην Επιτροπή Εκών το είχαμε συζητήσει, ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει πρόοδος και στην κοινοτική νομοθεσία γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο θέμα, δεν αφορά μόνο την Ισπανία, αλλά πολλά κράτη-μέλη. Τα δικαιώματα των καταναλωτών σε πολλά κράτη-μέλη. Απλά ε, έχει τριπλασιαστεί ίσω ο όγκο ε, των υποθέσεων στην Ισπανία σε σχέση με άλλε χώρε. Ο κύριο Τσίριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω όλα αυτά τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες, οι οποίοι θεωρώ ότι είπαν πράγματα με τα οποία συμφωνούμε όλοι και συμφωνώ και εγώ και η πολιτική ομάδα την οποία εκπροσωπώ. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε και μία πρακτική αξιολόγηση για το πόσο αποτελεσματικές είναι οι εργασίες εδώ της Επιτροπής μας, πώς μπορούμε δηλαδή να συμβάλλουμε έμπρακτα κι εμείς. Να ευχαριστήσω προφανώς αναφέροντες που είναι παρόντες εδώ, να επενθυμίσω ότι το ζήτημα αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας, και το θέμα αυτό δεν αφορά βέβαια μόνο την Ισπανία, αλλά και πολλές άλλες χώρες της ε, Ευρώπης. Πολλές φορές έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα με μία μάχη ανάμεσα στον Δαβίδ και τον Γολιάθ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συμβάλλουμε. Τέτοια φαινόμενα έχουμε προφανώς και στην Ιταλία. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε και σήμερα ότι ε, θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί πάρα πολύ στενά την εφαρμογή της συγκεκριμένης αυτής οδηγίας που έχει ως στόχο να προστατεύει τους καταναλωτές ενωπίων των τραπεζών. Θα πρέπει όμως να δούμε τι γίνεται και στο ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας, πώς δηλαδή εκδικάζει τις υποθέσεις αυτές και να καταφέρουμε τελικά να δούμε ποιες είναι οι ρήτρες εκείνες των συμβάσεων, μία προς μία, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν αθέμητες και καταχρηστικές. Νομίζω όμως ότι παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει και η απαραίτητη εκστρατεία ενημέρωσης των χρηστών και των καταναλωτών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι για μας το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η αναφορά αυτή από τεχνικής πλευράς τουλάχιστον θα μπορούσε να κλείσει διότι έχει παρέλθει και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σταματάμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στα φαινόμενα αυτά. Το αντίθετο. Το θέμα αυτό παραμένει ένα θέμα επί το οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα να μιλήσουμε εκ νέου για το ζήτημα αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση που δούμε βέβαια ότι οι διατάξεις της οδηγίας δεν τηρούνται. Η Σολεδάδ είναι η τελευταία. Και μετά θα κλείσω τον κατάλογο Το νομιτό Προσπαθήστε, Σολεδάδ, να είστε σύντομοι γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, σε σχέση με τα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι τελικά τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία αποφασίζουν ε, σε σχέση με την ερμηνεία της νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, και τελικά υπάρχει ασάφεια στα κράτη-μέλη και αβεβαιότητα. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει κάτι να πει γιατί ε, με την ασάφεια αυτή μάλλον η ΕΣΑΦ αυτή προκύπτει από την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, άρα αυτά πρέπει να αναφερθεί. Για την ε, προκειμένη περίπτωση, την περίπτωση τη Ισπανία, έχουμε και ένα επιπλέον πρόβλημα. Ότι δηλαδή η νομοθεσία για την υπόθηκα δάνεια δεν τηρεί ούτε τι διατάξει τη ισχύουσα νομοθεσία και τη σχετική οδηγία Ευρωπαϊκή Ένωση, εξού και κίνησε διαδικασία παραβάση Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη Ισπανία. Και όπω ε, είπε και ο συνάδελφο από το ΕΛΚ, δεν πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά, πρέπει να παραμείνει ανοιχτή γιατί αφορά όχι μόνο την Ισπανία, πολλέ χώρε. Απλά εμεί στην Ισπανία έχουμε και ένα παραπάνω πρόβλημα ότι είναι απαρχιωμένο ο σχετικό νόμο για τα ενυπόθηκα Δεν είναι και αυτό επέτρεψε την ύπαρξη αυτών των καταχρηστικών πρακτικών. Αυτή τη στιγμή γίνεται επεξεργασία μια νέα πρόταση νομοθετική. Ένα νομοσχέδιο είναι υποεκπώνηση και ελπίζουμε να είναι πιο σύγχρονο αυτό το νομοσχέδιο και να τηρεί και την ισχύουσα νομοθεσία. Βέβαια, στην περίπτωση συνολικά αυτών των ρητρών, στην Ισπανία έχουμε ένα πρόβλημα. Το έχουμε καταγγείλει και τον Οκτώβριο του 2015. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε και σχετική ετοιμιγορία. Και το είπε και ο αναφέρον. Η λύση που δόθηκε με το βασιλικό διάταγμα του 2017 δεν είναι αυτό είναι σαφές. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν όχι μόνο να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, αλλά και να στείλουμε στην Τράπεζα της Ισπανίας, για την Κεντρική Ισπανική Τράπεζα, μια επιστολή για να μας εξηγήσει τι μέτρα λαμβάνει επί του θέματος ώστε να εγγυάται τη μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία για τους καταναλωτές και στην Ισπανική κυβέρνηση πρέπει να στείλουμε μια επιστολή για να του πούμε ότι το θέμα το παρακολουθούμε και θέλουμε να σου πούμε τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία των καταναλωτών. Να λύσει με αποτελεσματικό γρήγορο τρόπο ε, κάτι το οποίο όλοι ε, θεωρούν ότι είναι αδικία. Είναι καταχρηστικές. τι πρακτικέ, το ξέρουμε. Άρα δεν είναι μόνο στο δικαστικό μέτωπο που πρέπει να εμείνουμε, αλλά γενικά πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα μια και πάντα. Να Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ξαναδώσω τον λόγο στον αναφέροντα, αφού ακούσαμε του συναδέλφου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ένα λεπτό όμω ή δυνατόν, για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Θέλω πραγματικά ειλικρινά να σας ευχαριστώ ε, για την προσοχή που δίνετε στην αναφορά που φορά πολλούς, όχι μόνο Ισπανούς ε, υπηκός, αλλά Ευρωπαίους πολίτες. Ε, εμείς οι πολίτες στην Ευρώπη βλέπουμε την τελευταία δυνατότητα που έχουμε στην διάθεσή μα, την τελευταία σανίδα σωτηρία στους κυβερνώντες στις χώρες μας, του εκλέγουμε. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει άλλη λύση και με του συντρόφου που συζητούμε πάντοτε λέμε λέμε θα έρθει η Ευρώπη και θα μας σώσει. Εκεί έχουμε να αποθέσει τι ελπίδε μας και ελπίζω να το κρατήσετε και αυτό κατά νου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, α προσπαθήσουμε να αποκριθούμε στα αιτήματά σας. Όπως είπε και ο κύριο Τσίριο πριν από λίγο, έχουμε εδώ πέρα μια κατάσταση Δαβίδ εναντίον Γολιάφα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε τη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σαφώ να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, καθότι αυτή τη στιγμή έχουμε εξελίξει διαδικασίε επί παραβάση. Κύριε Τσίριο, δεν είναι δυνατόν να να κλείσουμε την αναφορά τη στιγμή που τρέχουν ακόμα διαδικασίε επί παραβάση και περιμένουμε και μια απόφαση πολύ σύντομα μάλιστα. Πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά μέχρι να δούμε πώ θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίε επί παραβάση και πού θα καταλήξουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που είπε η Σολιντάντα, δηλαδή να έρθουμε σε επαφή με την Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας και να του θέσουμε κάποια ερωτήματα. Θυμάμαι την προηγούμενη Δευτέρα, όταν ήμουν στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το ζήτημα των συλλογικών προσφυγών όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αν τελικά αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει τώρα εν προκειμένου σε μια διαδικασία όπου έχουμε Δαβίδ και Γολιάθ. Ενδεχομένω λοιπόν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την διαιτησία, τη διαβου... την διαμεσολάβηση. Θα μπορούσε και αυτό να αποτελέσει έναν ελακτικό τρόπο επίλυση τη διαφορά αυτή. Και πραγματικά θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προ την Ισπανική Κεντρική Τράπεζα να διερευνήσει και τη δυνατότητα αυτή. Δεν είναι υποχρεωτικό το σύστημα που προβλέπεται, είναι προαιρετικό, αλλά δίδεται και αυτή η δυνατότητα τη διαμεσολάβηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν προκύπτουν τέτοια προβλήματα και όταν επιθυμούμε γρήγορα να βρούμε μία λύση. Α μην ξεχνάμε λοιπόν ότι εκκρεμούν αρκετέ προσφυγέ στα δικαστήρια. Συμφωνείτε με τη λύση αυτή. Πολύ ωραία και σα ευχαριστούμε πραγματικά που ήταν τόσο ακριβεί στην ε, παρουσίαση που κάνετε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το βιντεάκι το οποίο μα δείξατε. Σα ευχόμαστε καλή επιστροφή στην Ισπανία και αγοράστε και τίποτα βελγικά σοκολατάκια για να πάρετε μαζί σα. Και σίγουρα ο ήλιο που έχετε στην ε, Ισπανία είναι πολύ καλύτερο από ό,τι εδώ, αλλά οι σοκολάτες στο Βέλγιο είναι πολύ καλύτερες από τις Ισπανικές, θεωρώ. Λοιπόν, α περάσουμε στην επόμενη αναφορά, την υπαριθμόν 323 όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 2008 κάθετος 50 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη από τον Δήμο της Μαδρίτης και το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης. Ο αναφέρον είναι μαζί μας, είναι ο κύριος Αλεχάνδρος Σάντσες. Σας παρακαλώ πολύ, μην μιλάτε κι εσείς παράλληλα. Λοιπόν, Ας ακούσουμε τον αναφέροντα, τον κύριο Σάνσες. Κύριε Σάνσες, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μοιραστώ το χρόνο μου με την Ινέσα Βανέσα, τη συντρόφισσα που είναι δίπλα μου. Το 2011 το ΕΚΟ κατέθεσε αυτή την αναφορά γιατί το όζον και το διοξείδιο του αζότου ε, σημειώνουν υπερβάσει των οριακών του τιμών στη Μαδρίτη. Υπάρχει η ε, οδηγία 50 του 2008 η οποία παραβιάστηκε και κατατέθηκαν σχετικές αναφορές αλλά και φέτος το ίδιο. Και η Μανουέλα Καρμένα, η Δήμαρχος, ξεκίνησε στη Μαδρίτη μέτρα για την μείωση της ρήπανσης ε, και ιδίως σε ό,τι αφορά τη μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων ιδιωτική χρήση ε, που ε, είναι στην περιοχή Μαδρί Θεντράλ που έπρεπε να είναι υποτίθεται μια ζώνη χαμηλών εκπομπών και εκεί έχει περιορισμούς και στην κυκλοφορία από τις 30 Νοεμβρίου θα ισχύσουν. Αλλά στην κοινότητα της Μαδρίτης συνολικά δεν υπάρχει αυτή η αναθεώρηση. Υπάρχει το σχέδιο Μπλε Πλάσα το οποίο όμως δεν έχει εφαρμοστεί επαρκώς και δεν τηρούνται διατάξεις οδηγίας. Πάνω από 100.000 ε, κάτοικοι ε, όταν έχουμε ένα δήμο με 100.000 έχουμε προβλήματα, πάρα πολλά κολλήματα εφαρμόζονται, ώστε δεν μπορεί η κυβέρνηση Μαντρίτη να εφαρμόσει τα μέτρα και θέλουμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, ώστε να υπάρξει μια οριστική κατάληξη στη διαδικασία παραβάση κατά της Ισπανίας και στην ευρύτερη Μητροπολιτική της Μαδρίτης να ισχύσουν τα μέτρα τα οποία ισχύουν μόνο για το κέντρο. Ε, θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην Ινές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι υπάρχει το πρόβλημα της ρήπανσης. Ένα τεράστιο πρόβλημα, πάρα πολύ σημαντικό. Από το 2010 το βλέπουμε, όταν ξεκίνησε η νέα κυβέρνηση να, έχει, ε, να αναλάβει τα καθήκοντά της, ε, η δήμαρχος ε, της Μαδρίτης και εγώ μαζί είπαμε ότι τα αρχή μας προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και της αλλαγής του κλίματο, του κλίμα, καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Και έχουμε μέτρα όταν έχουμε εχμές ρήπανσης, μέτρα στρατηγικά επίσης. Άρα ε, και ε, κατά περίπτωση αλλά και στρατηγικά. Υπάρχει επίση μια επένδυση 500 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν αναλυφθεί διάφορα μέτρα, μεταξύ των οποίων ε, θέλω να τονίσω το σημείο 99 ε, της ε, εκθέση Κομισιόν που ζητά να υπάρχουν αυτές οι ζώνες χαμηλών εκπομπών. Αυτό γίνεται με τη Μαδρίτη Σεντράλ, αυτή την περιοχή του κέντρου της Μαδρίτης που από τα τέλη Νοεμβρίου θα αρχίσουν αυτοί οι περιορισμοί στην κυκλοφορία. Ζώνη λοιπόν χαμηλών εκπομπών, Μαδρίτη Σεντράλ. Είναι πολύ Θετικέ επιπτώσεις. Ε, θα είναι μικρό ο αντίκτυπο. Ε, ε, και σε ό,τι αφορά ιδίως τα πλέον ρηπογόνα οχήματα. και η διέλευση οχημάτων. Έχουμε συντονισμένη δράση μεταξύ της προηγούμενης και της νυν ισπανικής κυβέρνησης και της Κομισιόν. Μας δώσανε χρόνο ώστε το 2020 να έχουμε εφαρμόσει τους στόχους ε, και σε βάρος κάθε προγνωστικού ε, και παρά ε, την παρέμβαση από πλευράς των αρχών της Μαδρίτης που παρεμβαίνει στο έργο των τοπικών αρχών έχουμε καταφέρει πάντως κάποια πράγματα ήδη Θέλουμε να σεβαστούμε τα δικαιώματα των ενίκων αλλά και ε, ε, τη διανομή εμπορευμάτων κτλ. Θέλουμε απλά να περιορίσουμε ε, την κυκλοφορία των πλέον ρηπογόνων οχημάτων, αυτά τα οποία χρησιμοποιούν δίζελ και είναι πάνω από 10 χρόνια η ηλικία τους, ή παλιά οχήματα που κινούνται με βενζίνη και δεν έχουν και το σχετικό σήμα, την ετικέτα, όπως τη λέμε στην Ισπανία. Όπως συστήνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε λάβει αυτά τα μέτρα και νομίζω ότι καλό θα ήταν μια υπενθύμηση προς την κυβέρνηση και τις Ισπανικές Αρχές, ώστε να ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε σαφή αποτελεσματικά μέτρα, γιατί η θεμελιώδης αρχή είναι η προστασία, εναντί η προστασία της υγείας των πολιτών. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την Επιτροπή μαζί μας ε, και θα ήθελα να δώσω τον ε, Ντάνιελ Φερνάντες Κόμες ε, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες για την παρουσίαση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τη ρήπανση και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανησυχεί τα μάλα με την κατάσταση αυτή. Υπερεβάση συνεχής των οριακών τιμών που θεσπίζουν οι οδηγίες για την ποιότητα του αέρα για διάφορους ρήπους ατμοσφαιρικού στην περίπτωση της Μαδρίτης το βασικό πρόβλημα είναι το διοξίδιο του αζότου και επειδή αυτό το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης ε, είναι και βασική αιτία πρόωρων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο και μας ανησυχεί ακόμη περισσότερη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αποφάσισε να παρέμβει και να κινήσει διαδικασία παραβάση κατά των κρατών μελών εκείνων στα οποία παρατηρούνται συνεχείς ε, επίμονες παραβιάσεις και υπερβάσεις των οριακών τιμών που θεσπίζει οδηγία και εκεί όπου δεν λήφθηκαν ακόμη μέτρα ή σχέδια δράσης ώστε αυτές οι υπερβάσεις ε, να μειωθούν ή να πάψουν να υπάρχουν. Προτεραιότητα αρχικά έδωσε η Κομισιόν ε, σε συγκεκριμένες ουσίες. Ε, το διοξείδιο του αζότου είναι μια από αυτές τις ουσίες που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Μαδρίτη. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που πλήττονται ε, και από τις για τις οποίες έχει κινηθεί η δικασία παραβάση. Στις 30 Ιανουαρίου ο κύριος Βέλη, υπουργό Περιβάλλοντος, ε, κάλεσε διάφορα κράτη-μέλη για αυτό το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, εκεί όπου υπήρχαν ε, τα περισσότερα προβλήματα, έφτασε στις Βρυξέλλες για να γίνει μια συζήτηση και κατεπηγόντως να ληφθούν ε, αξιόπιστα και αποτελεσματικά μέτρα για να δοθεί ένα τέλος στο πρόβλημα αυτό που πλήττει τη δημοσία υγεία. Και να δώσουν και πληροφορίες ε, τα κράτη-μέλη για τα μέτρα τα οποία προτίθενται να λάβουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μετά από αυτή τη συνάντηση, τα κράτη-μέλη έστειλαν ε, τις ε, αιτήσεις πληροφορίες και η Ισπανική κυβέρνηση έστειλε τα μέτρα τα οποία προβλέπονταν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση της Μαδρίτης αλλά και στις άλλες ζώνες ε, και οικισμούς που περιλαμβάνονται στη διαδικασία παραβάσης που έχει κινηθεί. Μετά από ανάλυση των λόγω μέτρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην προσφύγει κατά της Ισπανίας στο δικαστήριο προς το παρόν για να δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστούν αυστηρά και εντός των προθεσμιών τα μέτρα που θεωρούμε ότι είναι ικανά να οδηγήσουν σε μείωση της, ε, ε, των επιπέδων του διοξιδίου του αζότου πριν το 2020 στη Μαδρίτη. Ελέγχουμε και παρακολουθούμε πάρα πολύ τους σύνεγγυς στην αυστηρή αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των μέτρων. Βλέπουμε κατά πόσο αποτελεσματικά ή όχι και αν διαπιστώσουμε ότι δεν εφαρμόζονται όπως είχαν αναγγελθεί τα μέτρα αυτά ή ότι δεν οδηγούν ε, στους ε, επιδιωκόμενους στόχους, ε, θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένω να καταφύγει στην, να προσφύγει στη δικαιοσύνη σε βάρο, κατά της Ισπανίας. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα δεν είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί για τις αποφάσεις των Ισπανικών δικαστηρίων δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Πενθυμίζω όμως ότι τα ισπανικά δικαστήρια υποχρεούνται και αυτά να εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις ε, που υπέχουν οι αρμόδιες αρχές ε, εφαρμόζονται, ότι τις λαμβάνουν ε, υπόψη τους δεόντως οι χώρες. Σολεδάβ, Καπεσόν Ρουή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που είναι εδώ. Η Μαδρίτη έχει ένα πρόβλημα ρήπανσης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί κανείς ε, να την αρνηθεί και αυτό φαίνεται και από τη δράση που έχει αναλάβει η Κομισιόν. Είναι ανοιχτή η διαδικασία παραβάση, ενδεχομένω να επιβληθούν και κυρώσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναφορά από το 2011 από την, όταν τότε ήταν το Λαϊκό Κόμμα στην κυβέρνηση που δεν είχε και ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό. Τώρα το Λαϊκό Κόμμα είναι αυτό που προτείνει να γίνει συζήτηση στην Επιτροπή Αναφορών για αυτό το ζήτημα. Μου κάνει λίγο έκπληξη αυτό. Ε, όταν η σημερινή κυβέρνηση ακριβώς λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν είναι λοιπόν φανεί όλα αυτά και δεν μας πείθουν ιδιαίτερα. Πρέπει να πω επίσης ότι η σημερινή ε, Δημαρχία της Μαδρίτης έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για να δοθεί λύση στο σοβαρό πολύ βέβαια αυτό πρόβλημα. Και χθες η κυβέρνηση της αυτόνομης περιφέρειας έκανε κάποιες ε, ανακοινώσεις ότι αφορά ακριβώς αυτό το σχέδιο το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει, προτίθεται να εφαρμόσει για τη Μαδρίδ Σεντράλ, περιορισμό κυκλοφορίας δηλαδή. Φαίνεται ότι το, η Δημαρχία κάνει ε, μάλλον η κυβέρνηση της Ισπανίας ε, κάνει και της και μα κάνει τις απαραίτητε προσπάθειες για την ε, αντιμετώπιση του προβλήματο στη Μαδρίτη. Η Άντζελα Βαλίνα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τη Σολεδάτ. Η Ισπανία έχει ένα πρόβλημα κατά την άποψή μου και όχι μόνο η Μαδρίτη γενικά. Γιατί στην, ε, στο φάκελο ε, δεν αναφέρεται μόνο η Μαδρίτη, αλλά και όλη η Ισπανία. Και αν δεν λυθεί το πρόβλημα, θα ε, πληρώσουμε τα πρόστιμα όλοι μας στην Ισπανία θα μας επιβληθούν καιρός. Και αυτό που μου φαίνεται επονίδιστο είναι τα προβλήματα στην Ισπανία να τα λύνουμε ή να αρχίσουν να μας απασχολούν με ψηφοφορίες μόνο και όχι με πολιτικές με επικεφαλαίο. Αν υπάρχει ένα σχέδιο, αν η Κομισιόν το παρακολουθεί και αν συμφωνεί με το πώς η κυβέρνηση της αυτονομίας ε, άλλου κόμματο, με άλλα αρχικά τέλο πάντων, δεν ε, εργάζεται προ το συμφέρον τη δημόσια υγεία των πολιτών, πραγματικά είναι κάτι το ακατανόητο, ιδίω από τη στιγμή που, παραλαμβάνω, αν υπάρξει πρόστιμο θα το πληρώσουμε όλοι μα με δημόσια χρήματα. Λυπούμε. Αν υπάρχει λύση πρέπει ε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί εγώ με τα δικά μου λεφτά κάνω ό,τι θέλω, όχι όμως με τα λεφτά τα δημόσια. Εκεί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θα μπορούσαν να είχαν λυθεί εδώ και χρόνια τα προβλήματα στη Μαδρίτη. Όπω είπε και αναφέρουσα, δεν επεδείχθη απαιτούμενη ευαισθησία κατά το παρελθόν, γιατί την τότε. Ε, τι τότε αρχέ δεν τι ένοιαζε. Τώρα που είναι η δαμόκλη σπάθη πάνω από το κεφάλι μα, πρέπει να το λύσουμε όμω το θέμα. Αλλά μετά τι γίνεται, βάζουν εμπόδια στο δρόμο και έχουμε την αυτόνομη κυβέρνηση να μην συνεργάζεται. Πραγματικά ε, είναι ε, τραγική αυτή η κατάσταση. Είναι σουρεαλιστικό αυτό που συμβαίνει. Θέλουμε να ε, εφαρμόσουμε πολιτικές υπέρ των πολιτών. Επιτέλους πια. Όχι ο ένας να στρέφεται ε, πολιτικός κατά του άλλου. Φυσικά και πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη η Κομισιόν και φυσικά και πρέπει να σταλεί επιστολή στην αυτόν περιφέρεια της Μαδρίτης. Να μας πούνε γιατί για ποιο λόγο δεν προχωρούν στην επίλυση ενός προβλήματος που αφορά την υγεία όλων των πολιτών. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ετωραγκάης. Συγγνώμη για την προσφορά. Όχι καλά τώρα προφέρετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω τους αναφέροντες, τον αναφέροντα και τη Δόνια Ινιές, την οποία την ξέρω από αυτή την Επιτροπή. που ξεκίνησε από την αντιπολίτευση και τώρα είναι μέλος ε, ε, του, Δημαρχείου, ε, του Δημοτικού Συμβουλίου με, και ασχολείται με τα θέματα του περιβάλλοντος. Συγχαρητήρια, Δόνια Ινιές. Αυτό το οποίο εγώ θα σχολιάσω, ελπίζω να σας κάνει να καταλάβετε λίγο ότι πόσο το αληθοφανές μπορεί να είναι και το μη αληθοφανές να είναι αληθοφανές. Όταν είχε κατατεθεί η αναφορά το 2011, όπως μας υπενθύμισε αναφέρουν. Μιλάει για την κοινότητα αυτών τη της Μαδρίτης αναφέρουν. Αλλά το Δημαρχείο ε, αναφέρατε, ε, ίσως εκ παραδρομής, τι κάνει η κυβέρνηση ε, της Μαδρίτης. Αυτό είναι το θέμα. Ε, που θέλω να σχολιάσω και την πολιτική που εστίασε και εστιάζει ε, στη, ε, στα δικαστήρια και στο πώς θα ρυθμιστούν ποιες θα είναι οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις, οι δρόμοι κτλ. Θέλω να δω τι γίνεται, όχι το τι έγινε όταν το 2011, αλλά τι γίνεται το 2017. Κάποιος δεν το παρέλειψε ε, να το πει. Το 2017 λοιπόν στο όζον και στο ε, διοξείδιο του αζότου είχαμε πέρβαση ε, στο 70% των σταθμών μέτρησης σε σχέση με τα προηγούμενα. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 η κυβέρνηση, θα το ξέρει πολύ καλά η κυρία Νιές, ενέκρινε το σχέδιο Α για την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή. Ένα σχέδιο το οποίο ε, αυτό που θα κάνει θα είναι να παραλύσει τη Μαδρίτη. Αυτό είναι ο στόχο ουσιαστικά. Ε, και φυσικά αυτό θα οδηγήσει, αν έχουμε συνέχεια κυκλοφορικέ συμφορίε, θα έχουμε και μεγαλύτερη ρήπανση. Όταν έχουμε αιχμές ρήπανσης ε, λόγω όζοντος ε, και διοξίδιο του αζότου πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση. Δεν γίνεται σωστή διαχείριση και το λένε και τα μέσα ενημέρωσης ε, και έχω και κάποια δημοσιεύματα. Και οι Μαδριλένοι ίδιοι είπαν ότι είναι αυτοσχεδιασμός πλήρης και χαοτικό αυτό το σύστημα το οποίο έχει προταθεί. Όταν οι πολίτες περίμεναν να δουν αν θα εφαρμοστεί μέτρο, μέτρο ή όχι, τους κορόιδεψε. Η κυβέρνηση και τα κοινωνικά δίκτυα και έχω εδώ ε, πάλι δημοσιεύματα. Υπήρχε ένα πρωτόκολλο το οποίο δέκα φορές ενεργοποιήθηκε και δημιούργησε δυσαρέσκεια ε, και μεγάλα προβλήματα. 15 από τις 24 σταθμούς μέτρησης που μετρούν το διοξίδιο του αζότου παρουσίασαν, σημείωσαν υπερβάσεις 40 ε, μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο. Άρα έχουμε πρόβλημα και στα μέτρα τα οποία προβλέπονται περιλαμβάνονται κάποια μέτρα έτσι κυκλοφορίας μέσω των φαναριών ε, που αυτό θα οδηγήσει σε 300% περισσότερα μποτιλιαρίσματα. Termino ya, 24 Οκτωβρίου 2018 άρχισε να ισχύει τότε ο νέος κανονισμός με περιορισμούς κυκλοφορίας, περιορισμό της στάθμευση των ιδιωτικών οχημάτων σε διάφορες περιοχές όπως το Madrid Central. Αυτό το διάταγμα δεν έχει κάποια υπόμνημα οικονομικό και απάντησε ε, η δημοτική κυβέρνηση και λέει να ε, δουν τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα. Μα είναι σκάνδαλο. Εμείς από το ΕΛΚ θέλουμε βέβαια να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, αλλά για να καταγγείλουμε αυτά που γίνονται τώρα στο Δημαρχείο. Αλλά όχι για το 2011, για το 2017, για τώρα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Επαναλαμβάνεστε το ξέρω ελπίζω, το ξέρετε ελπίζω. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνετε ακριβώ ό,τι έχει πει ο προηγούμενο συνάδελφο γι' αυτό σα παρακαλώ να μένετε, ε, να μένετε στα σημαντικά. Ε, εδώ η Άγγελα είπε ότι ε, συμφωνεί με τη Σολιδάθα, δεν χρειάζεται στη συνέχεια να επαναλάβει όλη την ιστορία, το ξέρω ότι είναι γυναικεία στρατηγική όμως ε, μπορεί να εφαρμοστεί και από τους άνδρες. Ε, ε, να ακούτε ο ένας τον άλλον, όμως δεν χρειάζεται να ξαναλέτε όλη την ιστορία από την αρχή, γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος. Βασελέση Εγώ όμως θέλω διαδικαστικό, λέει ο κύριος Σιντουργκάιθ. Κυρία Πρόεδρε, εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τι θέλετε να πείτε. Αλλά καταλάβετε, και κάτι. Τέσσερις συνάδελφοι παίρνουν το λόγο και καταφέρονται κατά τις δράσεις μιας συγκεκριμένης, ε, ενός συγκεκριμένου κόμματος. Τέσσερις μίλησαν κατά ενός και μένα ε, θέλετε να μου δώσετε ε, μία παρέμβαση ενώ έχετε δώσει τέσσερις παρεμβάσεις εναντίον μου. Και όχι, ολοκληρώνω. Μετά θα πάρετε το λόγο. Για λίγο σεβασμό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήρθε και ο κύριο από την Σκέρα Ρεπουμπλικά να καταλήγω να μα στήσει τέλο πάντων να δείχνουμε εμεί σεβασμό. Τέλο πάντων, στου συναδέλφου να πω. Εγώ έδωσα στοιχεία. Γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα. Όχι για λαϊκισμό και δημαγωγία. Ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρον να σας ακούω κύριε Ιτουργάης, αλλά όταν ο χρόνος περνάει και όλοι έχουμε έρθει εδώ για να ακούσουμε τους αναφέροντες και να βρούμε μια καλή λύση, αν έχετε μια καλή νέα συνεισφορά να κάνετε, κάντε την. Και ας είμαστε ε, λογικοί όμως. Ε, παρακαλώ κύριε, μας τελείωσε ο λόγος σε εσά. Ευχαριστώ, θέλω να ευχαριστώ και τους αναφέροντες και τον κύριο Σάντσεφ και το έργο που κάνουν είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να πούμε ένα βασικό νούμερο που το ξέχασε. Πέρα από τα μποτελιαρίσματα έχουμε πρόωρος θανάτους. 40.000 ε, το 2015 στην Ισπανία λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης ε, και υπάρχουν ε, συλλογικότητες που προτείνουν λύσεις όπως το Μαδρί Σεντράλ για να μειωθούν οι εκπομπές και να περιοριστεί η κυκλοφορία, έχουμε παρακόλληση αυτών των μέτρων από τους συντρόφους μας από το Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία από την κυβέρνηση τη αυτόνομη περιφέρεια τη Μαδρίτη, από την αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί έρχεται σε, ε, σε αντίθεση αυτό το μέτρο με την ανάγκη προστασία τη δημόσια υγεία. Γιατί η Βαλέθια, την Βαρκελόν, τη Μαδρίτη πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μα. Η δουλειά αυτή ε, την αναγνωρίζει και, το, ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κεντρική Κυβέρνηση που είναι από άλλο κόμμα, από το Σοσιαλιστικό και στη Μαδρίτη δεν ξέρω, το ξεχάσατε μάλλον, σας διέφυγε αυτό το στοιχείο, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε κατά 40% τη ρήπα κατά 40% τη ρήπα στη Μαδρίτη. Άρα αυτό που συμβαίνει ποιο είναι, ότι έχουμε παρακόλληση από την κυβέρνηση της, ε, ε, αυτών της περιφέρειας της Μαδρίτης, κατά των σχεδίων που συμφώνησαν η Μαδρίτη, η Κομισιόν και η Ισπανική κυβέρνηση. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο της δημόσιας υγείας, αλλά και των συμφερόντων της Ισπανίας, διότι για δική σας ευθύνη και για την επονίδιστη δική δική σας συμπεριφορά ε, θα πάμε ε, στα δικαστήρια πλέον. Θα μας πάει στα δικαστήρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και παρακαλώ να παραμείνει ανοιχτή αναφορά φυσικά και να στείλουμε αυτή την επιστολή που είπε η Σολεδά Διάχελα στην Ισπανία για να ζητήσουμε ε, να μας πει τι τι κάνει η κυβέρνηση εκεί και να πάψει να παρακολεί τα πράγματα και να δράσει προς όφελος των Ισπανών. Παρακαλώ, προσπαθήστε να σέβεστε όταν παίρνετε το λόγο τους αναφέροντες. Παρακαλώ, μην αρχίζουμε ε, εσωτερική ισπανική πολιτική στην καρδιά των ε, ευρωπαϊκών θεσμών. Δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Ήδη έχουμε ε, αρκετές ε, αρνητικέ θέσει από άλλε πλευρές. Εδώ είναι ένας ειρηνικό χώρο. Κυρία Μιράντα, έχετε τον λόγο και στη συνέχεια τελειώνει ο κατάλογος των ομιλητών και θα προχωρήσουμε. Παρακαλώ δείξτε ότι οι γυναίκε μπορούν να είναι συγκεκριμένε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Δόλα, καλωσορίζω του αναφέροντε γιατί έρχονται εδώ, γιατί πραγματικά υπάρχει αναλλακτική και αυτό θέλω να παρουσιάσουν. Όπω είπε η Πρόεδρο, οι γυναίκε έχουμε ε, μια διαφορετική αντιμετώπιση και προσέγγιση. Το κάναμε και με το ψήφισμα κατά του φασισμού Πεντρέμου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω επίση ε, και τι γυναίκε που διαπραγματεύτηκαν για όλα αυτά. Η Νέσ είναι η αρμόδια αυτό το θέμα και ξέρουμε ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Ξέρουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είπε πολύ ξεκάθαρα ότι πρέπει να γίνει σεβασμός και κοινωνικής νομοθεσίας, αυστηρή εφαρμογή. Εγώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δυστυχώς το Ισπανικό κράτος ήδη πληρώνει πρόστιμα στην περίπτωση ε, ε, των, της περιοχής Λαρίας πληρώνουμε και θα πληρώσουμε και άλλα, πολλά άλλα πρόστιμα. Εγώ κλείνω εδώ λέγοντας ότι στηρίζω ε, την ε, παραμονή της αναφοράς να παραμείνει ανοιχτή και πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε την κοινοτική νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Και τώρα θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στον, ε, στους αναφερόντες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα είναι απαραίτητη παρέμβαση της Κομισιόν. Πρέπει να παρακολουθεί αυστηρά ε, την κατάσταση και να βλέπει ότι η Ισπανία ε, τηρεί, ιδίω ε, στην περίπτωση της Μαδρίτης, όλα αυτά τα σχέδια. Επίσης, να σας καθησυχάσω. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν μοντελοποιηθεί από το Πολυτεχνείο και έχουμε αυτή την προθεσμία για το 2020. Από το 2018 έχουμε στοιχεία που δείχνουν σταθερή βελτίωση. Έχουμε αυτή την περιοχή χαμηλών εκπομπών που θα είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει την επιτεύξη των δεσμεύσεων και υποχρεώσεών μα. Για την επιστολή που λέτε να σταλεί στην Ισπανία, όπου θα απαιτείται όλε οι πλευρέ να τηρούν τι δικέ του υποχρεώσει, ε, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το Δήμο και πρέπει να σα πω ότι απέναντι στα προβλήματα τη κυκλοφορία, που ξέρετε ότι στι πόλει είναι πολύ σοβαρά αυτά τα προβλήματα, αλλά πέραν αυτού έχουμε τα προβλήματα που υπερτερούν τα προβλήματα της υγείας. Σήμερα στην Ελπαΐσα γίνεται λόγος για τις εχμές ρήπανσης ε, στη Μαδρίτη που ε, επηρεάζουν ε, τα παιδιά ε, και δημιουργούν προβλήματα υγείας, ιδίως για τα παιδιά. Αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει από όλε τι δίκες, αντί να ε, προχωρούν παρακολύοντας, να προχωρούν βοηθώντας ε, όλοι, όλες οι πλευρές. Σε συνεργασία και με την προηγούμενη Ισπανική κυβέρνηση, αλλά και τώρα, ακόμα με μεγαλύτερη ένταση, προχωρούμε γιατί οι στόχοι του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης γραμμίζονται πολύ με αυτά που κάνει η κοινότητα της Μαδρίτης αυτή τη στιγμή. Ωραία, αυτό το οποίο μας λέτε είναι ότι η κομματική πολιτική ε, και ότι η αναφορά αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια ομπρέλα για όλες ε, τις ε, κυβερνήσεις και πέρα από τα κόμματα. Η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας επί παραβάση θα αποστείλουμε μια επιστολή στις Ισπανικές Αρχές, ε, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης, αλλά και στην Κεντρική Κυβέρνηση. Τελεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Κεντρική Κυβέρνηση. Τελεία. Σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Ελβελπιστώ νέα είναι καλά οι αναφέροντες. Ευχαριστούμε που ήρθατε ε, στην, ε, στις Βρυξέλλες. Απολαύστε τον ήλιο. Ε, δεν είναι κάτι σύνηθες. Είναι η πολύ που μπορείτε να βιώσετε και, τους, και τις τέσσερις εποχές. Σεσίλια, μήπως θα έπρεπε να στείλουμε και μία επιστολή στην τοπική κυβέρνηση της Μαδρίτης γιατί αρμόδια δεν είναι η κεντρική κυβέρνηση, αλλά η αυτόνομη περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης. Μα αυτό είπα, και τα τρία επίπεδα θα πάρουν επιστολή. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα σημεία τη μερίδα διάταξη. Αποχωρήστε αθόρυβα και άμεσα, ώστε να συνεχίσουμε και με τα επόμενα σημεία. Το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη είναι το περιθμό 29, αναφορά 1226, Ιταλική αναφορά, επομένως διαφορετικό το στυλ αυτή τη φορά. Περιβαλλοντική Ένωση Κροτσεβία σχετικά με την περιβαλλοντική ρήπανση που έχει προκληθεί από πρώην βιομηχανική μονάδα και σταθμό απεξεργασία λιμάτων. Ο Ρομπέρτο Σενάτο είναι ο προσκεκλημένο μα που εκπροσωπεί τον αναφέροντα. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα για κάτι το οποίο συμβαίνει στο Ρέντε, στην πανεπιστημιακή πόλη του Ρέντε στην Καλαβρία. Λοιπόν, στη ζώνη αυτή, σε μία κτίνα 1,5 περίπου χιλιόμετρο, έχουμε δύο οικολογικέ βόμβε που υποβαθμίζουν την ζωή και την υγεία των πολιτών που κατοικούν σε αυτή την περιοχή όχι μόνο βέβαια τους κατοίκους, αλλά και τους κατοίκους που ζουν στις γειτονικέ περιοχές, στην ευρύτερη ουσιαστικά περιοχή. Έχουμε δύο οικολογικές βόμβες λοιπόν, το εργοστάσιο Λενιοκίμικα, καθώς επίσης και τη μονάδα καθαρισμού. Η Λενιοκίμικα ήταν ένα εργοστάσιο το οποίο αντλούσε τα νίνη από το ξύλο καστανιάς και το 2002 το εργοστάσιο αυτό σταμάτησε να λειτουργεί και μέσα σε 50 χρόνια λειτουργίας ξεφορτωνόταν με δύο τρόπους τελικά τα χημικά απόβλητά της ή τα απέριπτε στον ποταμό Κράτη, ο οποίος βρίσκεται εκεί δίπλα και ουσιαστικά καταστράφηκε οποιαδήποτε μορφή ζωής στον ποταμό αυτό ή τα τοποθετούσε σε υπόγειες, οκτώ υπόγειες μη στεγανές ε, λεκάνες, τις οποίες είχαν σκάψει μέσα στο έδαφος. Και όπως σας είπα δεν ήταν στεγανές. Δεν υφίσταται πλέον το εργοστάσιο αυτό, αλλά οι λεκάνες αυτές υφίστανται με όλα αυτά τα δηλητηριώδη απόβλητα, τρεις συγκεκριμένα γιατί οι πέντε στάφτηκαν κάτω από τη γη χωρίς να ακολουθήσουν εξιαντικά έργα. Οι υδροφόροι ορίζοντε έχουν μολυθεί πάρα πολύ και οι πυρογνώμονε που εξέτασαν την περιοχή θεωρούν ότι τα επίπεδα αλουμινίου, μαγκανίου, νικαλίου, σιδήρου υπερβαίνουν κατά πολύ τα ανώτατα όρια που προβλέπει ο νόμο. Αναφερόμαστε λοιπόν σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, σε μια πολύ επικίνδυνη ρήπανση. Το χειρότερο βέβαια πρόβλημα είναι ότι τα υγρά απόβλητα εξατμίζονται διαχέοντας στην ατμόσφαιρα μια ανυπόφορη δυσοδεία που φτάνει μέχρι το κέντρο της πόλης και αυτό υποβαθμίζει όχι μόνο την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και την ίδια την υγεία τους. Επίσης με τις ψηλές θερμοκρασίες εμφανίζονται φαινόμενα αυτανάφληξης και το καλοκαίρι προκύπτουν ακόμα και πυρκαγιές ξέσπασε μία πυρκαγιά κατά αυτόν τον τρόπο και κινητοποίησε πυροσβέστες για δύο ολόκληρες μέρες. Ο τοξικός καπνός από την πυρκαγιά κατέκλυσε το κέντρο της πόλης και ανάγκασε τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα μόνο ότι έκανε πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι του πρώην αυτού εργοστασίου έχουν ήδη πεθάνει από καρκίνο και τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση ογκολογικών παθήσεων. Βλέπουμε και πολύ σπάνιες νεοπλασίες ακόμα κυρίως στις οικογένειες που ζουν πολύ κοντά στις δύο αυτές μονάδες. Πολλά ήταν τα αιτήματα και κλήσει από περιβαλλοντικέ οργανώσει και από του κατοίκου που ζήτησαν να δημιουργηθεί ένα μητρό καταγραφή των καρκίνων. Και μετά από άοκνε προσπάθειε, το αρμόδιο δικαστήριο εξέδωσε μια διάταξη που ουσιαστικά ζητά από το Ιταλικό κράτο να προβεί σε εξυγίανση τη περιοχή, αλλά κάτι δεν έχει γίνει ακόμα πέρα από το πρόβλημα αυτό που έχει να κάνει με το εργοστάσιο λινιοκύμικα, έχουμε και το πρόβλημα που προκύπτει από τη μονάδα καθαρισμού. Η μονάδα αυτή δημιουργήθηκε στην περιοχή ενός πρώην αποτεφρωτή που έκλεισε το 1998. Οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της περιοχής αυτής παραπονιούνται και αυτοί για μια φόρητη δυσοσμία και το βράδυ και το πρωί και βέβαια αυτό εγείρει πάρα πολλές ανησυχίες για την υγεία των πολιτών και βέβαια πειράζει αυτό πάρα πολύ την ποιότητα ζωής όχι μόνο ο Δήμο ε, του ΡΕΝΤ έχει χαρακτηρίσει την περιοχή αυτή ω μια περιοχή που πρέπει να εξηγιανθεί και που θα πρέπει να μετατραπεί τελικά σε αστικό πάρκο, αλλά έχουμε και μια απόφαση του 2000 από την αρμόδια επιτροπή για τις περιβαλλοντικέ επίγουσες καταστάσεις τη περιοχή της Καλαμπρία, η οποία λέει ότι θα πρέπει να γίνει εξυγίανση, απορρίπανση τη περιοχή κάτι το οποίο δεν έχει γίνει βέβαια ακόμα. Και στι δύο λοιπόν περιπτώσει. Έχουμε απόβλητα τα οποία έχουν απορριφθεί στον ποταμό Κράτη και η έκθεση της Legambiente, της Οργάνωσης Προστασίας του Περιβάλλοντος Ιταλίας, έχει καταδείξει ότι στι εκβολέ του ποταμού Κράτη υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά τέτοια τοξικά απόβλητα. Δυστυχώ οι αρμόδιε αρχέ δεν έχουν προβεί σε καμία απορρίπανση και είναι πάρα πολύ σημαντικό τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει δράση προκειμένου να σταματήσει η αδιαφορία αυτή του ταλικού κράτου. Θέλουμε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα υγεία των πολιτών οι οποίοι ζουν κοντά στι δύο αυτέ μονάδε και να διαπιστωθεί επίσημα η παραβίαση τη Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία προκειμένου να εφαρμοστούν όλες αυτές οι αποφάσεις που έχουν ε, λάβει τα Ιταλικά δικαστήρια και προκειμένου να κληθούν οι αρμόδιες αρχές να εξηγιάνουν, να απορριπάνουν τις μολυσμένες αυτές περιοχές. Σας ευχαριστώ. Yeah. Και τώρα θα καλέσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής, Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει τον ε, λόγο, Μαρκό Γκασπαρινέτη, και παρακαλώ αν μπορείτε να επικεντρωθείτε στη διαδικασία επιπαραβάσης που υπάρχει στο ε, δικαστήριο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε μία συνήθη περίπτωση όπου σε μια πολύ φτωχή ζώνη ορισμένοι αποφάσισαν να πλουτίσουν προωθώντα ρηπαντικέ δραστηριότητε οι οποίε τώρα έχουν σταματήσει. Ξέρετε ότι έχουμε την οδηγία για τι βιομηχανικέ εκπομπέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προφανώ ισχύει και για την περιοχή αυτή. Εδώ έχουμε ένα εργοστάσιο που έκλεισε το 2002. Η εισαγγελία της περιοχής εκδίκασε και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου αυτού αλλά και τον αρμόδιο επίτροπο περιβαλλοντικής προστασίας οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή γιατί ακριβώς καταδικάστηκαν και στις δύο περιπτώσεις και οι δύο αυτοί εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες οι οποίες οδήγησαν σε περιβαλλοντική καταστροφή. Επομένως ανέλαβε δράση η Ιταλική δικαιοσύνη. Βλέπουμε ότι εκκρεμεί ακόμα η υπόθεση της που έχει ξεκινήσει ενώπιον της Αγγελίας όσον αφορά τον ε, αρμόδιο επίτροπο σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και όπως σας είπα, ο πρώην ιδιοκτήτης του εργοστασίου αυτού έχει ήδη καταδικαστεί ε, για λόγους περιβαλλοντικής καταστροφής. Θα πρέπει πέρα από τις ατομικές ευθύνες να δούμε πώς έχει όλη η διαδικασία σε τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και τι έχει γίνει σε τοπικό επίπεδο από τους ίδιους τους πολίτες και τις οργανώσεις των πολιτών. Βλέπουμε ξεκάθαρα εδώ πέρα ότι η κατάσταση δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς και ούτε έχουν δοθεί οι απαραίτητες ε, αποζημιώσεις. Αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε στην περιοχή του Τάραντο και ενός εργοστασίου που ε, υπάρχει στην περιοχή αυτή και στην συγκεκριμένη αυτή περιοχή δεν έχουν ληφθεί υπόψη αυτό το οποίο ονομάζει η Ιταλική νομοθεσία συγκεκριμένοι χώροι ε, κρατικού ενδιαφέροντος, εθνικού ενδιαφέροντος, στους οποίους θα πρέπει το Ιταλικό κράτος να προβεί σε απορρίπανση, σε εξηγεντικά μέτρα. Το Ιταλικό κράτο λοιπόν δεν έχει κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Εδώ και 16 χρόνια περιμένουν εξυγίανση οι πολίτε. Σε πιο τώρα υψηλό επίπεδο δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση πάλι, γιατί θεωρείται το ζήτημα αυτό από την Ιταλική πλευρά, θεωρείται το ζήτημα αυτό θα πρέπει να επιληθεί σε τοπικό επίπεδο, όπως ακριβώς είχε γίνει και στο, στην περιοχή του Τάραντο. Έχει προκύψει λοιπόν μια ενδιάμεση κατάσταση, την οποία θα πρέπει να εξολογήσουμε τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι η χρηματοδότηση για την εξυγίανση που δεν είναι εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε εδώ πέρα για τρει λεκάνε, οι οποίε θα πρέπει να στεγανοποιηθούν τροποντινά. Επομένω, οι αρμόδιες περιφερειακές δημόσιε αρχέ δεν καλούνται αυτή τη στιγμή να καταβάλουν ένα υπέρογκο ποσό. απορεί λοιπόν κανεί, για ποιο λόγο δεν έχει γίνει ακόμη η παρέμβαση αυτή. Τώρα, τι έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εσείς ε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μια συγκεκριμένη οδηγία που έχει να κάνει με τους υδροφόρους ορίζοντες και την προστασία τους και μετά την ε, πρώτη καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου και μετά τη δεύτερη καταδικαστική επίσης απόφαση του δικαστηρίου όπου ε, επιβλήθηκαν συγκεκριμένες κυρώσεις στην Ιταλία, εμεί περιμέναμε να ληφθεί περαιτέρω δράση από τι Ιταλικέ Αρχέ. Αναφέρομαι σε αποφάσει του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια. Όσον αφορά τι λεκάνες αυτές ε, στις οποίες έχουμε τα υγρά αυτά τοξικά απόβλητα, η απόφαση πρέπει να ληφθεί σαφώς σε τοπικό επίπεδο και να προχωρήσουν εκεί οι τοπικές αρχές τα απαραίτητα εξηγιαντικά μέτρα. Όπως ε, σα είπα όμω, σε επίπεδο Δήμου κοινότητα δεν έχει γίνει ακόμα κάποια παρέμβαση. Εμείς δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε όμω με τη διαδικασία επιπαραβάση, η οποία έχει να κάνει με τη μονάδα καθαρισμού, με τη μονάδα επεξεργασία λιμάτων, αλλά όχι με τι λεκάνε αυτέ, οι οποίε θα πρέπει να στεγανοποιηθούν και να σφραγιστούν. Αυτό, όπως σα είπα, αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και τα τοπικά δικαστήρια στην Ιταλία μιλάνε για περιβαλλοντική καταστροφή. Θεωρώ λοιπόν ότι με τη διαδικασία επιπαραβάση και τι καδικαστικέ αποφάσει που έχουν ληφθεί σε τοπικό επίπεδο, ενδεχομένω τα πράγματα να προχωρήσουν. Για πρώτη φορά με αντικατέστησε ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρότεινε αυτή, αντί να το κάνω εγώ, πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον, πώς θα πρέπει να κινηθούμε σταδιακά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που με αντικαταστήσατε στο ρόλο αυτό και που δείξατε αυτό το πολύ επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα έχετε το λόγο. Βλέπετε ότι εν προκειμένου η Επιτροπή μας δεν έχει μετατραπεί σε μια Ιταλική αρένα. Δεν είμαστε στη Βερόνα, αλλά στις Βρυξέλλες. Κύριε Τσίριο, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω και εγώ το λόγο για να ευχαριστήσω καταρχάς τους αναφέροντες που είναι εδώ και για να ευχαριστήσω όμως και το πολύ επικοδομητικό πνεύμα το οποίο δείχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ότι παρενέβη στα Ιταλικά. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε ότι όντω συμπάσχει, ότι όντω θέλει να συνεργαστεί για ένα πρόβλημα το οποίο πολύ εύκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί απλώ ένα τοπικό εθνικό πρόβλημα, κάτι που αφορά του άλλου και όχι την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε πολύ στενά το πώ εξελίσσονται τα πράγματα στην Ιταλία για μια υπόθεση η οποία είναι πολύ πλοκή πολύ, πολύ και πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα βήματα τα οποία θα κάνουμε, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει δικαστικέ διαδικασίε, όπω ακούσαμε, οι οποίε εκκρεμούν ακόμα. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, δεν θα πρέπει εμείς να επηρεάσουμε την όλη κατάσταση με μια πολιτική συζήτηση, θα πρέπει ως θεσμικό όργανο να επιτελέσουμε το έργο μας. Όπως είπε και η Πρόεδρος, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποιες εργασίες στεγανοποίησης έχουν λάβει χώρα ή όχι. Δηλαδή, τι όφιλε να κάνει η περιφέρεια, τι όφιλα να κάνουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για να αποκαταστήσουν μια τέτοια σημαντική περιβαλλοντική καταστροφή, τουλάχιστον για να μην συνεχιστεί αυτή η περιβαλλοντική καταστροφή. Νομίζω ότι ε, η δική μας η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην Καλαβρία και το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι προφανώς να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το πολύ, πολύπλοκο αυτό ζήτημα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να έχω άλλους ομιλητές ε, στον καταλογό μου. Θα ήθελε κάποιος, μήπως συνάδελφος, να λάβει το λόγο. Όχι, τότε καλώ τους αναφέροντες, ε, τον αναφέροντα μάλλον, ε, να ολοκληρώσει. Θα ήθελα να σχολιάσει κάτι ε, στο σχόλιο της Επιτροπής ή του κυρίου Τσίριο. Δύο λεπτά μέγιστος παρακαλώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποτανθούμε όντως στην περιφέρεια γιατί στην περιφέρεια της Καλαβρίας όταν προέκυψε αυτή η πυρκαγιά από περιφερεια της καλαβριας οταν προεκυψε αυτη η πυρκαγια απο αυταναφληξη Είχαμε τον επικεφαλή της περιφέρειας, ο οποίος ήρθε επί τόπου, ήμουνα και εγώ εκεί. Βλέπαμε ότι επί δύο ολόκληρες μέρες πυροσβέστες προσπαθούσαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά αυτή. Είδαμε ότι υπήρχε αυτός τοξικός καπνός που έφτασε μέχρι μέσα στα σπίτια των κατοίκων και τότε ο περιφερειάρχης μας έδωσε συγκεκριμένες υποσχέσεις. Δυστυχώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχει ξεκινήσει μια, ένα πινκ-πονγκ αν θέλετε αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πραγματικά ακριβώ που, που βρίσκονται οι ευθύνε. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ τον αναφέροντα που ήρθε από μακριά. Και τώρα θα ήθελα να ολοκληρώσω φυσικά και θα κρατήσουμε τη συγκεκριμένη αναφορά ανοιχτή. Η Επιτροπή ήδη μας βοήθησε πάρα πολύ, όμως αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω ε, προς την Επιτροπή είναι να παρακολουθεί αυστηρά όχι μόνο την Ιταλική συμμόρφωση ε, σχετικά με την οδηγία 91 2071 ε, αλλά επίσης ε, και την παραβίαση της οδηγίας ε, χιτά και βιομηχανικών αποβλήτων και πιστεύω ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε και σε αυτό εφόσον κάνετε μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη διαδικασία από πλευράς Κοινοβουλίου αποστέλλοντας ε, επιστολή στις, ε, Ιταλικές, ε, στις αρμόδιες Ιταλικές αρχές ούτως ώστε να αναλάβουν την αντίστοιχη δράση σε τοπικό επίπεδο. Μια επιστολή λοιπόν στην περιφέρεια της Καλάβρια ώστε να ενθαρρύνουμε και να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να συνεχίσει. Θα κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή και θα επανέλθουμε σε αυτήν αργότερα. Συμφωνούν όλοι με αυτό. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 30, το οποίο αφορά την παρακολούθηση τη διερευνητική επίσκεψη στη Μαδρίτη που έλαβε χώρα πέρσι τον ε, Μάιο υπό την ε, Root ε, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη ψυχολογικά επίσκεψη, επίσκεψη Έχουμε και τον εκπρόσωπο από την Αρχιεπισκοπή Λεμποπά. Πάτερ, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και θα ακούσουμε πρώτα τους αναφέροντες. Είναι η Άννα Κουέτο, Εσπεράνσα Ορνέδο και Ρουτ Άπλεμπι. Χαίρομαι ιδιαίτερω που είστε ανάμεσά μα για άλλη μια φορά. Έχετε έρθει και στο παρελθόν και τώρα θα ήθελα να σα δώσω το λόγο το πολύ 5 λεπτά ο καθένα. Which one starts? you're too humble. Just take the floor. Maybe, maybe... Είστε πολύ ταπεινοί. Ε, παρακαλώ ξεκινήστε. Ίσως η κυρία Ανακουέτο, την οποία αναφέρω και πρώτη. Τώρα να ξεκινήσω. Ναι, ναι ξεκινάω. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου ε, των ε, ενώσεων των θυμάτων που εκπροσωπώ, θα ήθελα να εκφράσω στην Επιτροπή σα ε, την απόγνωση, την εγκατάλειψη που νιώθουμε εμεί οι οικογένειε των αρπαγέντων παιδιών. Όποιοι μόνο έχουν ζήσει αυτή την κατάσταση, μπορεί κανεί να καταλάβει τι κενό νιώθηκαν στο να χάσει το παιδί του. Υπάρχει όμω και κάτι χειρότερο, την αβεβαιότητα, το ότι δεν ξέρουμε τι του συνέβη. Και είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι λόγω αυτού και εκτεθειμένοι στα μέσα ενημέρωσης Ελπίζουμε κάποια στιγμή ότι μπορεί να μας αναγνωρίσουν ίσως ε, αν μας δουν τα παιδιά μας, ίσως και στην τηλεόραση. Πολλά χρόνια ζήσαμε έχοντας την υποψία ότι κάτι έγινε με, το, με την απώλεια του παιδιού μας. Έχουμε ε, άδεια ε, φέρετρα από το 1993, το 2011, 18 χρόνια μετά παραμένει το κενοτάφιο σε ένα παιδί ή στο νεκροταφείο του Κάντιθ βλέπουμε αντίστοιχα τέσσερα, ε, πέντε φέρετρα λείπουν. Ε, είναι σκανδαλώδης ε, αυτή η κατάσταση νεογνά τα οποία δεν είχαν φτάσει να έχουν νομικό πρόσωπο για να καταγραφούν στα ληξιαρχεία. Μιλάμε τώρα ε, όχι για, το, τη μεταπολεμική εποχή ε, και μαζικού τάφους, ε, αλλά μιλάμε για δημοκρατική πλέον περίοδο. Όποτε προσπαθούμε να μιλήσουμε για μια τέτοια περίπτωση, που, για κάτι που έγινε στην δημοκρατική περίοδο, μας μιλάνε για την ιστορική μνήμη. και πάντα βρισκόμαστε σε ένα μετέωρο χώρο Πρόσφατα, ο ε, συνήγορο του πολίτη ε, μα είπε ότι 3.000 ε, ήταν οι καταγγελίε, δύο όμω δίκε έγιναν στη Μαδρίτη. Η Γενική Εισαγγελία έχει την εγκύκλιο 2 του 2012 που είναι αυτή που ρυθμίζει το πώς θα προχωρήσει η δικαιοσύνη. Εμείς λέμε πώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ε, ταυτοποίησης του θύματος. Ε, δεν μπορεί να αρχιοθετηθεί ε, η οδύνη των ε, θυμάτων. Υπάρχει μια θεσμική εμπλοκή. Μία μόνο απόφαση έχει ληφθεί μέχρι στιγμή. Η Ισπανική δικαιοσύνη δεν αναζητεί την βιολογική οικογένεια, ε, ούτε αναζητά τα χαμένα παιδιά. Υπάρχουν πολλαπλέ συστάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τα Ηνωμένα Έθνη. Η πραγματικότητα όμω των θυμάτων αυτή, τη μόνιμη, αυτού του μόνιμου εγκλήματο κατά ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δυστυχώ ε, ζούμε ακόμα αυτό το πρόβλημα. Στρεφόμαστε στον Οργανισμό ε, Θεμελιδών Δικαιωμάτων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να υπάρξει η Επιτροπή Έρευνα ε, για το δικαίωμα στην αλήθεια, στην επανόρθωση, για τη μνήμη των θυμάτων. Να ξεκαθαρίσουν όλε και να διαλευκανθούν όλε οι υποθέσει αρπαγή νεογνών. Ούτε παραγραφή υπάρχει, ούτε τιμωρησία μπορεί να υπάρχει, ούτε σύνορα μπορούν να υπάρχουν σε αυτέ τι περιπτώσει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κομισιόν που παρακολουθεί το θέμα για την ερευνητική επίσκεψη, γιατί πραγματικά πολύ πιστά μεταφέρατε ότι δημήφθη εκεί. Και σας ευχαριστούμε που έχετε ενημερώσει σχετικά και όλους τους ευρωβουλευτές. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Εδώ βλέπουμε τι έγινε ε, με το θέμα αυτό. Υπάρχει μια αίτηση ακύρωση ενώπιον του, του δικαστηρίου από την Αντουέθια Προβινθιάλ συγκεκριμένα. δεν ήταν δυνατό να ξεπεραστεί το πρόβλημα με την Αουντιένθια Προβινθιάλ. Καταγγέλουμε εδώ και χρόνια το θέμα ε, και θέλουμε να φτάσουμε στο ανώτατο δικαστήριο. Για πρώτη φορά στη μακρά δικαστική ιστορία ε, είναι ένα θέμα αυτό της αρπαγής ε, παιδιών που φτάνει στο ανώτατο δικαστήριο το οποίο μπορεί να καθορίσει την ομολογία Εδώ βλέπουμε την άποψη του ε, δικαστή Χωσέ Μαρία Μέντεθ Μπαρκίγιο, σε βάρο απόφαση του 12 και ανοίγει αυτή η δυνατότητα για ακύρωση ενώπιον του δικαστηρίου του ανώτατου και επίση ε, υπάρχει στήριξη του Γενικού Εισαγγελέα στη δική μα υπόθεση. Για πρώτη φορά στη δικαστική ιστορία τη Αουντέθια Προμηθιάλ τη Σουέλβα έχουμε έναν δικαστή που αποστασιοποιείται από την απόφαση τη Ολομέλεια του 12 και σε 34 φύλλα ε, αναφέρει τι πρέπει να γίνει ε, μιλάει για το νοδίνη των οικογενειών και αποφασίζει να βοηθήσει στην ε, πύληση του ζητήματος που έχει κολλήσει εδώ και έξι χρόνια και λέει ότι είναι θέμα συνείδησης, ε, στηρίζω μια υπόθεση που θεωρώ δίκαιη και την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. γίνεται λόγος για την παραγραφή, λέει ότι δεν μπορεί ε, να ε, παραγράφονται τέτοια αδικήματα και ζητείται να ξανανοίξει το θέμα και να υπάρχει ο δικός χάρτης. Ο εν λόγω δικαστής ε, στρέφεται κατά της Αντίενθια Προμηθιάλ και της απόφασης της και λέει μάλιστα ότι απορρίπτει ε, την ε, μεροληπτική ερμηνεία της Ολομέλειας. Θα κατατεθεί λοιπόν το θέμα στο Ανώτατο Δικαστήριο η δεύτερη προσφυγή ακύρωσης. και είναι η πρώτη φορά που υποτιθέμενα παραγραφέντα δικήματα θα ε, δικαστούν ε, στην Ισπανία. θα συνεχίσουμε και θα είμαστε όλο και πιο ισχυροί στην προσπάθειά μας να κερδίσουμε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ενδιαφέρον ε, να το βλέπουμε αυτό. Έχω ένα άρθρο συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη απόφαση της ε, απόφασης ένας ε, γυναικολόγος ε, κρίθηκε ένοχος από το ανώτατο δικαστήριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά ενισχύει την υπόθεσή σας. Ευχαριστώ λοιπόν που αναφέρατε και την δικαστική απόσταση, την απόφαση κυρία Άπελπη. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή την ε, συνάντηση. Πραγματικά είναι ε, χαρά μου και είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ. Ένα άλλο θέμα είναι να συζητήσουμε την υπόθεση γενικά και θα το κάνω αυτό χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες για την προσωπική μου υπόθεση, όμως είναι σημαντικό ότι καθώς είμαι θύμα το οποίο δεν ζει στην Ισπανία. Αρκετές από τις συστάσεις σας ήταν, ε, αφορούσαν και εμένα και θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε αυτά τα θέματα τώρα. Η σύστασή σας, υπαριθμών 7, είναι ξεκάθαρη σχετικά με το ποια ποιες αρχές είναι υπεύθυνε ε, για την έρευνα δεν έχω καμία απόδειξη ότι από την αναφορά και έπειτα έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή και πραγματικά δυσκολεύομαι να βρω τον οποιονδήποτε ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη διεξαγωγής έρευνας ε, πέραν ε, ημών. Οπότε είναι σημαντικό για μένα διότι ε, στην Europol στη σελίδα 10 αναφέρεται η υπόθεσή μου και η Ισπανική το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ισπανίας δεν γνωρίζει την υπόθεσή μου και αυτό διότι η Βρετανική αστυνομία διεξήγαγε έρευνα. Όλα αυτά είναι όμως ψευδή και είναι εξοργιστικό ως θύμα να διαβάζω κάτι τέτοιο. Ύστερα από 6,5 χρόνια βρίσκομαι ακόμα στην ίδια κατάσταση, είναι ασυγχώρετο. Η υπόθεσή μου έχει περάσει όλο το ισπανικό ε, ε, δικαστικό σύστημα, ακόμα και το συνταγματικό δικαστήριο και κάθε απόφαση έχει επικυρωθεί από τον δημόσιο εισαγγελέα. Οπότε, πώ τολμούν να λένε ότι δεν γνωρίζουν την υπόθεσή μου. ...κατά τέτοιο είναι ασυγχώρητο. Συγγνώμη, είμαι ιδιαίτερα συναισθηματική, διότι είναι ασυγχώρητο. Έχω αγωνιστεί για την υπόθεσή μου για πάρα πολλά χρόνια. Ε, χρήματα, αγάπη, χρόνος και το μόνο που μου δίνουν ως απάντηση είναι ότι δεν ξέρουν την υπόθεση μου. Η Βρετανική αστυνομία μου είπε ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αυτά ήταν τα λόγια τους. Ότι είναι σαν τον ταχυδρόμο. Ότι ο ρόλος τους με την Ιντερπολ ήταν απλά να παραδώσουν τα έγγραφά μου, την υπόθεσή μου, τίποτα άλλο. Και το ξανακούω αυτό. Πού βρίσκομαι λοιπόν. Η Βρετανική αστυνομία λέει ότι δεν μπορεί να παρέμβει ε, στο δικαστικό σύστημα μιας άλλης χώρας. Η, ε, ο, ο εισαγγελέας της ε, Ισπανίας λέει ότι δεν, ξέρει τίποτα για μένα, οπότε είμαι χαμένη μέσα σε αυτό το χάος όπου κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Ούτε και, η δική μου η χώρα θα πρέπει να αναλάβει ευθύνη έχω εξαλείψει όλες μου τις δυνατότητες στην Ισπανία διότι έχω πάει σε κάθε δικαστήριο που θα μπορούσα και όλο αυτό τον καιρό κανένας δεν μου μίλησε. Ούτε ένας. Και δεν μπορώ να καταλάβω το πώς μια υπόθεση μπορεί να πάει στα δικαστήρια με ε, ζήτησα να καταθέσω σε ε, δικαστή, όμως πάντοτε μου αρνούνται αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω ποιος λαμβάνει την απόφαση. Δεν ξέρω. Πέραν της ε, νομοθεσίας που έχω σε ένα έγγραφο, το οποίο λαμβάνω κάθε φορά που η υπόθεση μου κλείνει. Η θέση μου λοιπόν είναι ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι δεν υπάρχει ενεργή έρευνα και επειδή δεν μπορούν να παρέμβουν. Τι να κάνω λοιπόν. Η υπόθεση μου μπορεί να ξανανοίξει μονάχα στην Ισπανία σε περίπτωση που βρεθούν νέα στοιχεία. Πώς θα βρω νέα στοιχεία όταν δεν ε, ανοίγεται η υπόθεση, ότι δεν όταν δεν υπάρχει ενεργή υπόθεση. Αναφέρεστε επίσης το ότι θα πρέπει να βρεθεί το τι έχει συμβεί ασχέτως της ε, νομικής βιωσιμότητας. Στην υπόθεση μου αλλά και στην υπόθεση άλλων αναφερόντων εδώ όλο αυτό έχει αποτύχει διότι τα έγγραφά μου όλα έχουν γίνει νομικά. Κανένας δεν έχει ελέγξει όμως το τι έχει συμβεί. Μου δόθηκε μια ε, άδεια να θάψω το παιδί μου που δεν έχει υπογραφεί. Απαράδεκτο. Ζήτησα έλεγχο των ε, δεκτυλικών αποτιμάτων. Ε, τίποτα. Δεν έγινε. Όλες οι υποθέσεις που έχω υπόψη μου έχουν τεράστια ποσότητα εγγράφων, τα οποία όμως κανένας δεν εξετάζει και ήταν ενθαρρυντικό να διαβάσω στην έκθεση ότι το βάρος της δικαστικής διαδικασίας θα πρέπει να αφαιρεθεί από το θύμα. Όμως τίποτα δεν συμβαίνει. Ε, θα μπορούσατε, παρακαλώ, να ολοκληρώσετε, λέει η πρόεδρος. Εκτός μικροφώνου. λόγω του, της διεθνούς διάστασης της υπόθεσης μου και επειδή η Ιντερπόλ εξετάζει ε, μια διασυνοριακή υπόθεση. Η υπόθεση μου πήγε στην Ιντερπόλ, δεν έγινε τίποτα. Ζήτησα να μιλήσω μαζί τους, δεν μίλησα με κανέναν. Δεν θέλω να κλείσω αρνητικά όμως. Η Επιτροπή Αναφορών όμως με έχει υποστηρίξει πάρα πολύ, δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Η θέση μου αυτή τη στιγμή είναι ότι πραγματικά ε, πιέζω την ε, τοπική μου αστυνομία να λάβει χρηματοδότηση από το Home Office. Ε, χρειάστηκε ένας χρόνος, εδώ και ένα μήνα ζητάω ενημέρωση. Με ενημέρωσαν την Τετάρτη, μόλις είπα ότι θα έρθω εδώ και μόνο χάρη στην Επιτροπή Αναφορών, αν κάτι προχωράει, είναι χάρη στην Επιτροπή Αναφορών. Νιώθω ευάλωτη διότι από τον Μάρτιο του 19 η χώρα μου έλαβε μια πολύ άσχημη απόφαση και η οργή η οποία βλέπετε είναι τεράστια. Υπάρχουν νέες υποθέσεις ε, στη Μεγάλη Βρετανία. Έρχονται σε μένα να ζητήσουν βοήθεια. Εργάζομαι. Πρέπει να φροντίσω τα παιδιά μου, να βγάλω βόρτα το σκύλο ε, και ταυτόχρονα πρέπει να ακούσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχω μια Ισπανίδα κυρία με Βρετανίδα μητέρα, προσπαθούμε να τη βρούμε. Εγώ το κάνω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, ζητάει η αναφέρουσα. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι ε, έρχονται άνθρωποι σε μένα που ζητούν βοήθεια, αλλά πού πάω εγώ. Καταλαβαίνω, λέει η πρόεδρος. Ε, έχουμε συνέστηση για αυτό το οποίο περνάτε. Τώρα θα ήθελα να στραφώ στους εκπροσώπους των ε, οργανώσεων θυμάτων ε, που ε, συμμετείχαν στην νέα νομοθετική πρόταση. Έχουμε δει κάποια κινητικότητα στην Ισπανία και θα χαρώ να ακούσω για αυτό από την κυρία Σολιδάθ και, την, και τον κύριο Παρέκο. Τρία λεπτά στον καθένα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, καλημερίζω όλα τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση Σήμερα κλείνει ένα χρόνο από τη δημοσίευση τη έκθεση τη Δημοτική Αποστολή και των Συστάσεων. Εξαιρετική έκθεση που συμπίπτει με την νομοθετική πρωτοβουλία τη ΘΕΑΚΟΑ, δηλαδή τη κρατική συντονίστρια που στηρίζει ε, την υπόθεση Αργεντινή για πρόταση νόμου για τα αρπαγέντα παιδιά ε, στην Ισπανία. Κάτι το οποίο βασίζεται στι αρχέ των ΗΕ για το δικαίωμα στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αποζημίωση και για να μην επαναληφθούν φαινόμενα. Και συμπεριλαμβάνει τη συστάση τη έκθεση Επιτροπή Αναφορά. Το 2016-2017 η δική μα η Ένωση, τα παιδιά που έχουν αρπαγεί είναι τα δικά μου παιδιά, ε, συνεισέφερε στην τροποποίηση του νόμου 33-2013 στην Ναβάρα και στην τροποποίηση του νόμου Δημοκρατική Μνήμη ε, τη Βαλένθια με στόχο τα θύματα αρπαγή παιδιών να συμπεριληφθούν στι νομοθεσίε των αυτόνομων περιφερειών. Ε, τα δύο νομοσχέδια έγιναν δεκτά 29 Ιουνίου και 19 Οκτωβρίου του 2017. Με αυτές τις ε, εμπειρίες λοιπόν και όταν αρχίσαμε πλέον να βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα πλαίσιο ε, κρατικό για τις ε, διάφορες νομοθετικές διαστάσεις των αυτονομιών λόγω της ιδιαιτερότητας του εγκλήματος αυτού σε σχέση με άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι διερμηνείς διαμαρτύρονται γιατί μιλάτε πολύ γρήγορα. Μήπως θα μπορούσατε λίγο να πάτε πιο αργά για να μπορεί να μεταφράζετε αυτό που λέτε. Lo siento. Ναι, λυπούμε. Έλεγα ότι με αυτές τις εμπειρίες από τις αυτόνομες περιφέρειες συνειδητοποιήσαμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κρατικό πλαίσιο σε αυτές τις ε, περιφερειακές νομοθετικές διατάξεις λόγω της ιδιαιτερότητας του εγκλήματος αυτού σε σχέση με άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Συνήθως ο προορισμός ε, των νεογνών τα οποία τα άρπαζαν ε, ήταν μακρινός σε σχέση με τον τόπο γέννησης η δράση σε επίπεδο αυτόνομη περιφέρεια, αν δεν υπάρχει διασύνδεση με τι άλλε κοινότητε, δεν διευκολύνει το να μπορέσουν να βρουν τα παιδιά του οι ούτε τα παιδιά αυτά που σήμερα είναι ενήλικες να ανακτήσουν τη χαμένη του ταυτότητα, γιατί είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται οι μεν και οι δε σε τελείως διαφορετικά σημεία της Ισπανικής επικράτειας ε, και επομένω, ε, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν ε, στις νομοθεσίες των αυτόνομων περιφερειών πρέπει να συνοδεύονται από ομοιογενείς μηχανισμού. Θα πρέπει επίση να δημιουργηθούν διαφορετικοί φορεί και κρατικά, ε, κρατικοί μηχανισμοί ώστε να μπορεί να ερευνάται αυτό το έγκλημα σε όλο το κράτος με συντονισμένο τρόπο. Όταν ξεκαθαριστεί αυτή η αναγκαιότητα μάλλον αφού το ξεκαθαρίσαμε αυτό, ε, στραφήκαμε στην Θεάκουα σε, σε αυτή την, στο ε, φορέα συντονισμού, όπου συμμετέχουμε και εργαζόμαστε από τότε που συγκροτήθηκε το 2012. Είναι ένας οργανισμός που έχει ήδη μακρά πορεία στον αγώνα πράσπισης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλές δράσεις έχει αναλάβει, μεταξύ των οποίων η πρόταση νομοσχεδίου για τα παγέντα νεογνά, την προσπογράφουν όλα τα πολιτικά κόμματα. 25 Σεπτεμβρίου κατατέθηκε την Τρίτη, δηλαδή πριν δύο μέρες, 20 Νοεμβρίου, η Σοσιαλιστική Ομάδα την κατέθεσε στην Ολομέλη για να ληφθεί υπόψη και εγκρίθηκε ομόφωνα ε, η διεκπαιρέωσή της. Είναι κάτι ιστορικό πραγματικά. Πόσα λεπτά μου μένουν. Ναι, γι' αυτό το λόγο ε, και για μας αυτή η πρόταση, αυτό το νομοσχέδιο που θα ε, προωθηθεί ε, και με την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών αλλά και της κυβέρνησης ε, είναι το σημαντικότερο βήμα που έχει γίνει από νομοθετικής πλευράς. Υπάρχουν ε, πλέον τα εργαλεία ώστε το κράτος επιτέλους να εκπληρώσει την υποχρέωσή του που είναι να διερευνήσει την αλήθεια, να δικαιώσει τα, δίκτυμα, τα θύματα, να τους δώσει αποζημίωση, να δικαστούν οι θήτε και να μην ξαναεπαναληφθεί ποτέ αυτό το τρομερό έγκλημα. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από την Επιτροπή σας να κάνει μια ανακοίνωση για την ανάγκη να δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατόν η έγκριση αυτού του νομοσχεδίου για τα αρπαγέντα νεογνά στο Ισπανικό κράτο πριν το τέλο τη ε, θητεία αυτή. Σα ευχαριστούμε. Thank you very much and I didn't want to interrupt it. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα να διακόψω διότι ήταν πολύ ενδιαφέρον και ήξερα που θα το πάτε. Πριν από δύο μέρες είχαμε αυτή την ομόφωνη υιοθέτηση το οποίο αποτελεί ε, ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα από το Ισπανικό Κογκρέσο και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφό σας για άλλα τρία λεπτά. Καλημέρα και εγώ θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου όπως η ε, προλαλή σας ε, για την ε, πρόσκληση μας που να συμμετέχουμε στην συνάντηση αυτή και σε συνέχεια της επισκεψής σας στη Μαδρίτη 22 23 Μαΐου ε, έχουν κατατεθεί συστάσεις 23 Νοεμβρίου του 2017. Έκτοτε, ε, δηλαδή από το Νοέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018, οι Ισπανικές αρχές ούτε σε ό,τι αφορά την αναγνώριση, ούτε σε ό,τι αφορά τη διαρρήνωση του κλίματος έχουν σημειώσει πρόοδο κατά τη δικτατορία του Φράγκο και για τα πρώτα χρόνια της μεταπόλησης, της ε, δημοκρατικής μετάβασης. από τότε που άλλαξε η κυβέρνηση τον Ιούνιο, έχουν γίνει κάποια άτολμα, αλλά τέλος πάντων απαραίτητα βήματα πρόοδου για να αναγνωριστούν αυτά τα εγκλήματα. Το και η Σολεδά Δλούκε, η προλαλήσασα. Την Τρίτη η Ολομέλεια ε, εξέτασε αυτό το νομοσχέδιο και εγκρίθηκε ομόφωνα η ε, έναρξη της ε, όλης αυτής ε, διαδικασίας. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε κάποιες βασικές αρχές της πρώτας περιλαμβάνουν και συστάσεις της δικής σας επιτροπής. Για πρώτη φορά εγγυάται αυτό το νομοσχέδιο τα δικαιώματα για τα θύματα αρπαγής παιδιών. Αναγνωρίζεται επίσης το δικαίωμα στην αλήθεια δικαιοσύνη, την επανόρδωση και τιμή επανάληψη με διάφορα μέτρα. Παραδείγματος χάρη θα έχουν τα θύματα πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και δημόσια και ιδιωτικά, παραδείγματο χάρη τα αρχεία των κλινικών νοσοκομείων της Καθολικής Εκκλησίας. Επίσης θα γίνουν εκταφές με βάση και μάλλον με το αίτημα και του Υπουργείου Δικαιοσύνη και όχι από τα θύματα πλέον. Θα υπάρχει νομική, ψυχολογική και ιατρική ε, μέρημνα και υποστήριξη και μερτικές εκστρατείες από τις δημόσια για να μην επαναληφθεί ποτέ αυτό το έγκλημα στο μέλλον. Ναι. Αναγνωρίζεται η συνθήκη του θύματο ε, για αυτού που έπληξαν από αυτό το έγκλημα. Είναι ένα έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα. Η Ισπανία αρχίζει επίση να εφαρμόζει τι συστάσει των Μένων Εθνών, ιδίω ε, σε ό,τι αφορά την ε, δικαιοσύνη για την μεταβατική αυτή περίοδο και τι αρχέ του διεθνού δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για πρώτη φορά πλέον αναγνωρίζεται αυτό το καθεστώς θύματος ε, για, όσους, ε, για, τις απαγές παιδιών και για την περίοδο της δικτατορίας και για μετά. Ε, υπάρχει λοιπόν μια νέα δυναμική η οποία δημιουργείται Θέλουμε λοιπόν να δημιουργηθεί και μια ειδική εισαγγελία, είναι αυτό κάτι που αναφέρεται και στο νομοσχέδιο, που θα ερευνά και Θέλουμε επίσης να υπάρχει μια μονάδα έρευνας της δικαστικής αστυνομίας και μια κρατική επιτροπή για το δικαίωμα στην ταυτότητα. Και για να μπορέσουν να εργαστούν αυτοί οι οργανισμοί θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων για απογραφή και βάση εθνικού DNA. Με αυτό το σύστημα επίσης εγγυημένη συμμετοχή των θυμάτων μέσω των εκπροσώπων του και υπάρχει μεγάλη στήριξη από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ε, υπέρασπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγώ λοιπόν ζητώ να ζητηθεί από την Ισπανική κυβέρνηση να εγκρίνει αυτό το νομοσχέδιο και βέβαια η πλειονότητα των συστάσεων ε, να ε, εφαρμοστούν, γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα παρά λίγε και αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήδη λέμε ότι είχαμε μια υπέροχη συνεργασία μεταξύ των αναφερόντων ε, της Επιτροπής μας και η απόδειξη αποτελεί αυτό εδώ το έγγραφο ότι το Ευρωπαϊκό Κογκρέσο και η ε, διαδικασία που έχει ξεκινήσει αναφέρεται στην Επιτροπή μας και τα όσα έχουμε κάνει για να το μελετήσουμε. Το θέμα αυτό δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι κάτι το οποίο αφορά τους πάντες ή αφορά την δικαιοσύνη, αφορά την ανθρωπιά. Είναι μία υποχρέωση για τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας των πολιτών ε, να ε, υψώσουν τις φωνές τους, να ανοίξουν τα αρχεία, να ε, μιλήσουν. Μόνο η ελευθερία θα μας απελευθερώσει και δεν είναι λάθος το να αφήσουμε την αλήθεια να λάμψει. Τώρα να στραφώ στην εκπρόσωπο της Επιτροπής, την Ζωή Ζακυλιάδου και σας καλώ να εξηγήσετε την θέση της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω την συμπαράστασή μου για τα όσα είπαν τα θύματα. Σίγουρα είναι δύσκολο να παίρνεις το λόγο ύστερα από τέτοιες ιστορίες. Μαζί με ε, την συνάδελφο της Επιτροπής εξετάσαμε τις αναφορές των θυμάτων όσον αφορά τα νομικά εργαλεία. Εμείς εξετάσαμε ε, στο θέμα στο πλαίσιο της οδηγίας κατά του τράφικινγκ διότι κάποιες από τις ε, ε, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε τέτοια ανησυχία. Ε, επικοινωνήσαμε με τους ε, αναφέροντες και τους είπαμε ότι τα χέρια μας είναι δεμένα, ότι οι υπόθεσεις αυτές είναι πριν την οδηγία και πριν από την αρμοδιότητά μας να εξετάσουμε τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτό όσον αφορά την οδηγία κατά του τράφικινγκ. Ίσως για το ε, μέλλον θα θέλαμε να τονίσουμε ότι μία από τις προτεραιότητες μας είναι να ε, λήξουμε την ατιμορρησία για τους διακινητές και όλους όσους βοηθούν και υποφελούνται από το έργο τους. Ε, ως Επιτροπή είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό το θέμα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συνάδελφό μου η οποία παρακολουθεί την οδηγία για τα θύματα. Ονομάζομαι Καταλίνα Ανιέσκα Είμαι από την Κοινική Διεύθυνση δικαιοσύνη και θα ήθελα να αναφερθώ στην οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων. Η οδηγία αυτή είναι μια διαδικαστική οδηγία και γι' αυτό το λόγο είναι εφαρμοστέα και σε εγκλήματα τα οποία έλαβαν χώρα στο παρελθόν και πριν από την έναρξη σε ισχύ του εργαλείου αυτού δεδομένου ότι οι ε, ποινικέ διαδικασίες όπως και οι έρευνες λαμβάνουν ε, χώρα ύστερα από την έναρξη σε ισχύ της οδηγίας. Οπότε η συγκεκριμένη οδηγία εγκρίθηκε το 2012, άρχισε ε, να ισχύει το 15 Νοεμβρίου το 2015, οπότε τα δικαιώματα των θυμάτων υπάγονται σε αυτή την ε, οδηγία και είναι εφαρμοστέα σε όλες τις ποινικέ έρευνες ε, που γίνονται από 15 Νοεμβρίου του 2015 και έπειτα τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα υποστήριξης ε, από εμπειρογνώμονα, από γενικές υπηρεσίες, το δικαίωμα σε προστασία, το δικαίωμα ε, πρόσβασης σε πληροφορίες. Ε, υπάρχουν και άλλα γενικά δικαιώματα τα οποία αφορούν ε, θύματα και είναι δεσμευτικά για όλους ε, όσους έρχονται σε επαφή με τα θύματα κατά τη διαδικασία των ε, νομικών διαδικασιών. Επίσης, έρευνες, τα θύματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, αξιοπρέπεια, χωρίς διακρίσεις και με βάση τις μεμονωμένες ανάγκες των θυμάτων στην Επιτροπή δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με μεμονωμένες υποθέσεις ε, ιδιαίτερως όσον αφορούν ε, την εξέβρεση δεδομένων. Όλα αυτά ε, επαφίονται στις εθνικές δικαστικές αρχές, όμως η Επιτροπή παρακολουθεί το πώς τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την οδηγία δικαιωμάτων των θυμάτων και αυτή τη στιγμή ελέγχουμε την εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών και της Ισπανίας. Το 2019 η Επιτροπή θα εκδώσει μία αναφορά σχετικά με το πώς όλα τα κράτη-μέλη και η Ισπανία λοιπόν έχουν διασφαλίσει ότι ώστε τα θύματα μπορούν να βασιστούν στα δικαιώματά τους στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που το διευκρινίσατε. αν εφαρμοστεί αυτό ε, από τα κράτη-μέλη και εκτελεστεί ορθώς από τα κράτη-μέλη θα βοηθήσει ιδιαίτερος και θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Είναι λοιπόν ενθαρρυντικό για τους αναφέροντες ε, για να προσπαθήσουν να ερευνήσουν και να δουν αν η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων ε, μπορεί να βοηθήσει ε, διότι ισχύει σε όλες τις ε, ποινικέ υποθέσεις για την πρόσβαση στην πληροφόρηση για παράδειγμα. Η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι ένα σημαντικό στοιχείο διότι λαμβάνοντας τις σωστές πληροφορίες ήδη νιώθεις μία ενθάρρυνση το να μην ξέρεις απολύτως τίποτα είναι το χειρότερο. Θα ήθελα τώρα να περάσω στους συναδέλφους ε, και αρχικά θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, Jude Garland. Ευχαριστώ Σίλια. Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας την υπομονή σα, διότι αυτή είναι ίσως η τελευταία φορά που θα μου δίνετε η δυνατότητα να μιλήσω για αυτές τις αναφορές και εργαζόμαστε πάνω σε αυτές τις αναφορές ε, καθ' όλη τη διάρκεια τη ε, θητείας του Κοινοβουλίου και λόγω του ε, Brexit δεν θα μπορέσει να προχωρήσει αυτό. Δεν το περίμενα αυτό. Είναι, μια, είναι και στην ομάδα μα έχουμε εργαστεί στενά με τους αναφέροντες αλλά και με άλλους και πιστεύω ότι το ανανεωτικό είναι ότι παρόλο που υπάρχει ε, πόνος ε, και νιώθουν ότι βρίσκονται ε, στη μέση του πουθενά, τα πράγματα παρόλα αυτά κινούνται και αυτό είναι καλό να το αναφέρουμε ένα χρόνο μετά. Όπως γνωρίζετε ήταν μία δύσκολη και αποστολή όπου συναντήσαμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και η έκθεση την οποία ε, ε, ψηφίσαμε αντικατοπτρίζει ε, το συνολικό συνέστημα της αποστολής και αντικατοπτρίζει ταυτόχρονα τα, τις απαιτήσει των αναφερόντων προς αυτό το κοινοβούλιο και αυτό το οποίο ακούσαμε λοιπόν σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι δηλαδή έχουμε, ε, έχουμε κάνει μια μεγάλη διαφορά ως Επιτροπή Αναφορών και πραγματικά είχαμε μια άμεση επιρροή σε αυτό το θέμα και αυτό το καταλάβαμε όταν πρωτοξεκινήσαμε όπου και θεωρούσαμε ότι είναι μια χαμένη υπόθεση γονείς, παιδιά που ψάχνουν συγγενείς, γονείς, αδέρφια νιώθαμε ε, σαν και αυτούς ότι βρισκόμαστε στο πουθενά. Ε, όμως η Επιτροπή αυτή, η Επιτροπή Αναφορών, ε, προσέφερε ελπίδα, ενότητα σε αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάτι πολύ ισχυρό συμβαίνει και ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και μετά την θητεία μου και τη θητεία αυτού του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν χάρηκα ιδιαιτέρως που την Τρίτη έλαβα ένα mail από την Μαδρίτη όπου μου έλεγαν ότι ε, το Ισπανικό Κοινοβούλιο ομοφόνος είχε ψηφίσει την νομοθεσία για τα κλεμμένα βρέφη. Η πρόταση περιελάμβανε επίσης ε, τις περισσότερες συστάσεις μας. Φαίνεται ε, ότι έχουμε επηρεάσει και η συζήτηση που είχαμε με την Επιτροπή Δικαιοσύνης του Κοινοβουλίου όπου βουλευτές έλεγαν μεταξύ τους το πόσο ντροπιαστικό ήταν για τους ίδιους ότι χρειάστηκε αποστολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάει στη, στο Μαδρί, στη Μαδρίτη για να μπορέσει να ε, προχωρήσει λιγάκι τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των κομμάτων Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίζουμε, οπότε εντάχει ήθελα να τονίσω μερικά από τα βασικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε αυτό το νομοθετικό κείμενο. Πρώτον, καλεί όλους, να, να χρησιμοποιηθούν όλοι οι πόροι για την ε, εξέβρεση της αλήθειας σχετικά με την κλοπή βρεφών στην Ισπανία από τις 17 Ιουλίου το ε, 36. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι η συζήτηση αυτή ήταν πολύ έντονη συναισθηματικά και έπρεπε να δούμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κληρονομιά του Ισπανικού εμφυλίου. Αναγνωρίζοντας όμως ότι η έναρξη είναι ο εμφύλιος της Ισπανίας, είναι σημαντικό για τα θύματα για, ε, όσον αφορά αυτήν την αναζήτηση. Όλοι λένε ό,τι έχει πει ο Νέλσον Μαντέλα σχετικά με το μακρύ χέρι της δικαιοσύνης ε, και ισχύει και εδώ. Επίσης, το δικαίωμα στην αλήθεια σημαίνει ότι τα θύματα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα, έγγραφα ε, νοσοκομείων, ε, νεκροταφείων και δημιουργεί μια εθνική βάση DNA για την εξέβρεση ανθρώπων Αναγνωρίζει στα θύματα ότι έχουν ε, το δικαίωμα δωρεάν ε, παροχής ε, ιατρικής, ψυχολογικής περίθαλψης και το βάρος εξέβρεσης της αλήθειας δεν υπάρχει άλλο πια στο θύμα. Όλοι μας έχουν, τα θύματα έχουν μουδιάσει από την αναζήτηση της αλήθειας. Είναι λοιπόν σημαντικό το ότι ψηφίστηκε την Τρίτη, όμως ε, τώρα οι βουλευτές, οι νομοθέτες ε, γνωρίζουμε ότι έτσι ξεκινά η διαδικασία και εμείς όπως Επιτροπή Αναφορών βοηθήσαμε ούτω ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε λοιπόν να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να εθαρρύνουμε το Κοινοβούλιο της Ισπανίας να προχωρήσει ως το τέρμα και οι προτάσεις αυτές, οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ούτως ώστε να δοθούν απτά δικαιώματα στους αναφέροντες ε, που εκπροσωπούμε. Επίσης, σε περιφερειακό επίπεδο στην Ισπανία θα πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν πιο γρήγορα, το οποίο επίσης είναι πιο αισιόδοξο. Τα τελευταία χρόνια ήρθαμε σε επαφή με διάφορα μέρη με τον Αρχιεπίσκοπο Λεμπεπον, πρέσβη του Βατικανού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βοήθειά του ήταν πολύ θετική, ούτως ώστε να βρούμε ε, λύσεις ε, σχετικά με τις ανησυχίες μας ε, που γύραμε στη Μαδρίτη σχετικά με την πρόσβαση στα εκκλησιαστικά αρχεία η Επιτροπή επιβεβαίωσε λοιπόν ότι τα εκκλησιαστικά αρχεία υπάγονται στον κανονισμό ε, ε, GDPR και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ο καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτά όταν θέλει να βρει δεδομένα για τον εαυτό του ε, σε εκκλησιαστικά αρχεία. Από την επισκοπική διάσκεψη είχαμε επιβεβαίωση ότι τα εκκλησιαστικά αρχεία θα δοθούν ε, ελεύθερα μαζί με δημόσια αρχεία, ώστε να έχουμε ε, πληροφορίες ε, και δεδομένα τα οποία έχει κρατήσει η Εκκλησία. Θα χαρώ να δω να προχωρά αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τις ε, μονάδες της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Μας βοήθησε ιδιαιτέρως. Ε, είχαμε την ε, οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων και υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις που έχουν αρχιοθετηθεί αλλά δεν έχουν κλείσει διότι θεώρησαν ότι ότι οι συμμετέχοντες έχουν πεθάνει επειδή λείπαν πληροφορίες. Όμως όλες οι υποθέσεις που έχουν αρχιοθετηθεί ισχύουν στο πλαίσιο το, της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων και θα πρέπει να δούμε δράση από τις ισπανικές αρχές ούτω ώστε η οδηγία αυτή να εφαρμοστεί πλήρως στο πλαίσιο αυτών των υποθέσεων. Και θα ήθελα επίσης να αναγνωρίσω ότι οι αναφέροντες έχουν αυτοοργανωθεί και οδήγησαν στη δημιουργία ενός δικτύου ονόματι We are looking for you, σε ψάχνουμε, το οποίο ε, δείχνει ότι υπάρχουν και άλλα διεθνή παραδείγματα και θα πρέπει να δούμε το πώς θα υποστηρίξουμε αυτό το δίκτυο. Είναι αυτοοργανωμένο, όμως είναι ευάλωτοι, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν υποστήριξη και εμείς ως Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν το τι μπορούμε να κάνουμε και επίσης θα ήθελα να ευχαριστώσω τον Αντώνιο Αλόνσο Αλόνσο από το Εθνικό Κέντρο INTCF που ήταν συνεχώς σε επαφή μαζί μου έστελνε mail από την Ισπανία, μου εξηγούσε πώς προχωράει η κατάσταση και αυτό είναι σημαντικό. Έχοντας πει λοιπόν όλα αυτά και επειδή είναι η τελευταία μου ευκαιρία να μιλήσω, θεωρώ ότι πολλά έχουν προχωρήσει, όμως ακόμα έχουν πολλά να γίνουν. Ως Επιτροπή λοιπόν αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι οι αναφορές αυτές να παραμείνουν ανοιχτές, διότι ρίχνοντας φως στο τι συμβαίνει δημιουργούμε ένα πλαίσιο ούτω ώστε να συνεχιστεί η αναζήτηση της αλήθειας στην Ισπανία και καλό τον πρόεδρο του ε, Ισπανικού Κοινοβουλίου αλλά και τον επικεφαλής ε, της Επιτροπής Δικαιοσύνης ε, του Κοινοβουλίου της Ισπανίας ότι θα χαρούμε να κλείσουμε αυτές τις αναφορές και να δώσουμε ε, την τον έλεγχο της μάχης στους ε, Ισπανούς, ε, ε, στους Ισπανούς βουλευτές. Όμως θα πρέπει να δούμε την απόφαση της Τρίτης να περνά και να εφαρμόζεται σε όλο το δικοστικό σύστημα της Ισπανίας. Θα σταματήσω εδώ είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία όχι μονάχα σε αυτή την επιτροπή και με τους αναφέροντες και με τους συναδέλφους στην Μαδρίτη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό τόσο στην Ισπανία όσο και εκτός της Ισπανίας και μόνο με αυτή την δημόσια συζήτηση θα μπορέσουμε να λάβουμε απαντήσεις για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ε, το βάρος αυτής της αναζήτησης ε, που νόμιζαν ότι πραγματικά ψάχνουν σε τα νερά και μπορέσαμε λοιπόν να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ Τζούντα. Ως επικεφαλής Επιτροπής Αναφορών θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω ολόθερμα για όλη την εργασία που κάνετε για το ζήτημα αυτό. Πραγματικά αποτελείται υπόδειγμα. Υπόδειγμα μιας αξιοπρεπούς μεθόδου εργασίας και πραγματικά το επίτευγμα είναι καταπληκτικό. Και νομίζω ότι ε, σε προσωπικό επίπεδο θα πρέπει πάντα να μπορείτε να συνδυάζετε αυτό το πάθος σας, την αποφασιστικότητά σας και την ενσυναίσθηση που δείχνετε προς τους άλλους. Και πάντα λάμπει και υπερτερεί στο τέλος η αλήθεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ εξ ονόματος Επιτροπής μας. Κάντε εξαιρετική δουλειά. Ευθύνομαι τώρα στους υπόλοιπους συναδέλφους που ήταν παρόντες στην διερευνητική αυτή αποστολή και που θέλουν να πάρουν το λόγο. Η Καρμπεσόν Ρίθ πρώτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν. Δράτω με τις ευκαιρίες για να εκφράσω και εγώ την αλληλεγγύη μου προς τους αναφέροντες και για να αναγνωρίσω και το ρόλο της Επιτροπής Αναφορών, το ρόλο που είχε και εξακολουθεί να έχει σε αυτό το θέμα και μπόρεσε έτσι να δώσει δημοσιότητα σε αυτό το θέμα και να επηρεάσει και τη ε, δράση της Ισπανικής Κυβέρνησης. Θέλω να ευχαριστήσω την Τζούντ ε, που πραγματικά έχει καταθέσει σημαντικές συστάσεις στο πλαίσιο της έκθεσης, και αυτή τη αντιπροσωπεία με υποδειγματικό τρόπο και εν γέννη θέλω να σε ευχαριστήσω ε, συνολικά για το έργο στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναφορών. Μεγάλη ευαισθησία έχεις δείξει, ίσως είναι η τελευταία φορά που σε ακούμε εδώ, δυστυχώς ε, λόγω Brexit και της κατάστασης που γνωρίζουμε, όμως Ήθελα να πω, Τζουντ, ότι έπρεπε να σε ευχαριστήσω όλο ειλικρινώ, ιδίω δε για την προκειμένη αυτή περίπτωση. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει αλλαγή. Υπάρχει μία πρόταση, ένα νομοσχέδιο που δρομολογήθηκε και θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μίλησε πολύ ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη οδηγία για τα θύματα. Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα αλλάζουν, χωρί βέβαια να μπορούμε ακόμα να θεωρήσουμε ότι πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά. Θα έλεγα λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή και να ζητήσουμε, αφού ζητήσουμε να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, ε, να γίνει μια κατεπίγουσα συζήτηση στο πλαίσιο της Ισπανικής Βουλής, ε, ώστε να δρομολογηθεί αυτή η εξέταση και η έκριση του νομοσχεδίου. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαριά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, οι αναφορές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές Καταρχάς να συγχαρώ τους αναφέροντες που είχαν το κουράγιο να έρθουν εδώ στην Ευρωβουλή εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό για να θέσουν το ζήτημα, το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα και από πολιτικής και ιστορικής απόψεως της αρπαγής ε, παιδιών κατά τη διάρκεια του δικτατορικού καθεστώτος του Φράγκο αλλά και διαδικασιών που συνεχίστηκαν και μετά ε, όταν ε, άρχισε να υπάρχει αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ε, και το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάθεση νόμου στην Ισπανική Βουλή για το θέμα αυτό νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιτυχία. Να συγχαρώ τη Τζούντιθ και τους άλλους ε, συναδέλφους που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί διότι πήραμε αυτή την υπόθεση όταν ξεκίνησε εδώ και τα πράγματα ήταν και λίγο τα πνεύματα οξυμένα και συζητήσαμε αυτή την υπόθεση σε βάθος. Δεύτερον, είχαμε την απόφαση να στείλουμε μία fact-finding mission για να δει πώς έχει το θέμα Τρίτον, έγινε συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό και επομένως νομίζω ότι αυτή η πρακτική που ακολουθήσαμε σε συνδυασμό με τη μεγάλη δημοσιότητα έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα μπορεί να είναι και ένας οδηγός για το πώς σε μεγάλα σημαντικά θέματα πρέπει να ενεργεί η Επιτροπή αυτή. Γνωρίζετε ότι ασχολούμαι με το θέμα της Επιτροπής Αναφορών από το 1992-93 γράφοντας άρθρα για το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι η περίπτωση αυτή είναι κλασική. Βέβαια θα περίμενα να δω και άλλους συναδέλφους Ισπανούς εδώ, διότι θυμόσαστε ότι την πρώτη φορά που το συζητήσαμε είχαμε εκπροσώπηση όλων των συναδέλφων από την Ισπανία και επίσης όταν υπάρχει μια ισπανική ε, αναφορά είναι γεμάτη εδώ η αίθουσα από Ισπανούς συναδέλφους. Δεν ξέρω τώρα, καθώς ολοκληρώνεται θετικά αυτή η εξέλιξη, δεν βλέπω εδώ που θα έπρεπε να έρθουν και οι ίδιοι να επικροτούν αν θέλετε αυτή την κατάληξη τη θετική διότι νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα όλων και όχι μόνο μερικών. Σε κάθε περίπτωση να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, να δούμε πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω. Εύχομαι αυτό το νομοσχέδιο να ψηφιστεί στη Βουλή της ε, Ισπανίας και από εκεί και πέρα να μείνει ανοιχτό διότι τώρα είναι πλέον το θέμα των ίδιων των πολιτών και των αρχών της Ισπανίας να αρχίσει αυτός ο έλεγχος για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και εμείς σαν Επιτροπή να είμαστε ανοιχτοί για να παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα το οποίο νομίζω έχει συγκλονίσει όλη την Ευρώπη και πολύ περισσότερο βεβαίως την Ισπανία γιατί είναι ένα ανθρώπινο ζήτημα αλλά και με ιστορικές διαστάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία αυτού του ζητήματος. Μίλησαν κάποιοι για τις ανεπάρκειες της ισπανικής δικαιοσύνης ε, ή της Ισπανίας εν γέννη και εγώ δεν θα επιμείνω γιατί κάποιοι μπορεί να βρουν ε, ε, στα λόγια μου κακοπροαίρετες προθέσεις γι' αυτό δεν θέλω να το κάνω γι' αυτό θα μιλήσω μόνο για τα θετικά τελικά περνάω στα ισπανικά τώρα τελικά λέω έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο το περιμέναμε και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό νέο, ένα μεγάλο νέο. Όμως ε, υπάρχει ένα προβληματάκι που φαντάζομαι ότι θα λυθεί. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, τέλος πάντων. Η αναζήτηση ταυτότητας στην προκειμένη περίπτωση από φιλοσοφικής πλευράς αυτό μου φαίνεται δύσκολο. Όλοι θέλουμε να έχουμε μια ταυτότητα. Αυτοί που ξυλοκοπήθηκαν, που ε, ε, φυλακίστηκαν, ε, που απήχθησαν. Ε, εντάξει, κάπως πρέπει να το διατυπώσουμε, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά η αναγνώριση της καταγωγής για πολλά αρπαγέντα παιδιά θα δώσει κάτι στην ταυτότητα που έχουν τώρα. Αλλά Ελπίζω να έχουν ήδη ταυτότητα που την έχουμε όλοι μας και ακόμα και οι μητέρες που έχουν περάσει από αυτό το γολγοθά έχουν μια ταυτότητα όπως και να το κάνουμε. Τώρα το κείμενο λέει ότι ήταν πάνω από 30.000 τα παιδιά. Μα όχι, ήταν πάρα πολύ περισσότερα. 200.000 μπορεί και να ήταν, μην πω 300.000. Ε. Λοιπόν, πρέπει να το ξαναδούμε αυτό λίγο, έτσι. Επίσης, Κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, αυτό που ε, έκανε η Τζούντ ε, και είπε σε ό,τι αφορά τα αρχαία της Εκκλησίας. Εγώ τι κατάλαβα, Τζούντ, αν μπορείς να με ακούσεις, όταν πήγαμε Μαδρίτη, αν κατάλαβα καλά τότε από αυτά που μας είπανε οι εκπρόσωποι, οι επίσημοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, ήταν ότι τα αρχεία της Εκκλησίας εξαρτώνταν, ότι αυτοί δεν κάναν τίποτα, γιατί εξαρτώνταν από την κάθε επισκοπή ή άλλη θρησκευτική συνάθρηση ή φορέα. Αυτό θέτει ένα ενδιαφέρον ζήτημα μεν και πρέπει να το δούμε. Τώρα, μπορεί να γελάσετε τώρα λίγο μαζί μου, αλλά εμένα ξέρετε τι με ανησυχεί τώρα. Ότι είναι ένα πάρα πολύ μακροσκελές κείμενο αυτό. Δεν είχαμε τίποτα και τώρα έχουμε ένα πάρα πολύ μακροσκελές κείμενο, πολύ καλό σε, πολλές του, σε πολλά του σημεία, αλλά Δημιουργούνται δύο πράγματα που δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχουν. Δημιουργείται η κρατική επιτροπή για το δικαίωμα στην ταυτότητα. Δημιουργείται η ειδική εισαγγελία για τα αρπαγέντα ε, βρέφη, παιδιά κτλ. Πολλά και διάφορα μπορούμε να πούμε. Ή ότι η συγκεκριμενοποίηση από κρυστάλλους όλων αυτών θα μπορούσε να γίνει όταν εμείς θα έχουμε πεθάνει πια ε, και αυτό που πρέπει να γίνει νομίζω είναι να πάνε γρήγορα τα πράγματα. Δεύτερο, να προχωρήσουν τα πράγματα αλλά με συντονισμένο τρόπο για να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Θα το δούμε αυτό όμω φαντάζομαι. Θα το δούμε όπω εξελίσσεται η νομοθετική διαδικασία. Άρα, έχουμε εμπιστοσύνη, όμως ε, προειδοποιώ για αυτά τα προβλήματα. Πολύ καταπληκτικό αυτό το έγγραφο ε, που το εγκρίνουμε μεν, αλλά υπάρχουν προβλήματα, όλα αυτά, η δικαιοσύνη, η επανόρθωση κτλ, κτλ. Καλά και άγια. Αλλά συγκεκριμένα τι κάνουμε. Επομένως, και εδώ ολοκληρώνω σιγά σιγά κι εγώ. Τι ήθελα να πω. Α. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη διαδικασία, στα αγγλικά τώρα μιλάμε, και ότι πρέπει να είμαστε ανοίκτοι κτλ. κτλ για αυτή την αναφορά και ότι πρέπει να ζητήσουμε από την Ισπανική κυβέρνηση, ίσως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κατά βασά πιθανότητα τέλο πάντων του αρμόδιους φορείς, ώστε Τέλο πάντων, νομίζω στην επιστολή μα πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ. Είμαστε ικανοποιημένοι. Χαιρόμαστε ε, που υπάρχει μια πρώτη αντίδραση στις ανησυχίες μας και μια ανταπόκριση μετά την επισκέψή μας στην ε, Ισπανία. Δεν είναι έτσι, αλλά έτσι το ερμηνεύω εγώ τέλος πάντων. Ένα ε, πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, όμως ταυτόχρονα θα θέλαμε να παραμείνουμε ενήμεροι τι; διότι Μα ενισχύει τόσο πολύ το θέμα. Είναι τόσο σημαντικό για μα που θα θέλαμε πάρα πολύ να θα ενήμεροι για τα θετικά βήματα που γίνονται με την επίτευξη των στόχων. Αυτό νομίζω θα ήταν μια καλή αντίδραση εκ μέρους μας ε, που θα βοηθήσει να γίνει κατανοητό ότι δεν επαναπαυόμαστε, όχι, Θέλουμε να παρακολουθούμε τα πράγματα συνεχίζουν, προχωρούν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχω κάποιον άλλον ομιλητή. Απευθύνομαι τώρα πάλι στους αναφέροντες. Θα ήθελα ένα από εσά να πάρει το λόγο για δύο λεπτά απλώς για να αντιδράσει γρήγορα στα όσα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίας αυτής. ποιο θέλει να πάρει το λόγο. Ας ε, ολοκληρώσουμε όπως ξεκινήσαμε. Sí, Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε για κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε μόνο δύο δυνατότητες. Έχουμε το σημείο της τεκμηρίωσης και τις ε, δοκιμές, τα τεστ, τις εξετάσεις. Ε, και τα δύο προχωρούν. Εδώ έχουμε μια έκθεση από το Εθνικό Ινστιτούτο Ταξικολογίας και δικαστικών Ερευνών. Ο γιος μου όμως έχει ταφεί σε δύο διαφορετικά μέρη. Και στην έκθεση αυτή εγώ δεν μπορώ να ταυτοποιήσω τη δική μου περίπτωση ούτε όλες τις άλλες ε, περιπτώσεις εκταφών που έγιναν εκταφές ε, σε φέρτερα που δεν είχαν μέσα σωρό που αποκαλύφθηκε ίσως ότι το φθορός δεν ανήκε στην οικογένεια. Εγώ ούτε ένα στοιχείο δεν αναγνωρίζω από καμία σπανική οικογένεια εδώ. Δεν υπάρχει καμία αναφορά, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχει σε αυτή την έκθεση καμία αναφορά. Επειδή λοιπόν ε, είναι ελεγχόμενο το θέμα της τεκμηρίωσης, οι μόνες ε, ε, δυνατότητες που έχουμε πλέον εμείς είναι να αποδείξουμε ότι τα παιδιά μας δεν πέθαναν και δεν έχουν ταφεί εκεί που λένε ότι τα θάψανε. Πραγματικά ζητώ να υπάρξει μια ευθύνη σε σχέση με τις εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή σας. Αυτό εδώ είναι κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία έχετε πάρει από το έτος 1991 και για τα παιδιά μόνο. Ε, απλά. Δεν υπάρχει όμως κάτι που να αφορά τις αρπαγές των ε, παιδιών. Τυχαία το βρήκα αυτό το έγγραφο και το είδα τυχαία και το λέω όσα αναφέρουσα, ως μητέρα που ψάχνει το γιο της που έχει ταφεί σε δύο διαφορετικά σημεία. Ευχαριστώ. Thank you very much Σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την ε, διαλλακτική στάση την οποία δείξατε και πραγματικά πετύχει κανείς ε, να δείξει ιδιαίτερα θα, ιδιαίτερο θάρρο για να πάρει το λόγο όταν υποφέρει ιδίω τόσο πολύ για κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που πήρατε το λόγο, που ήρθατε εδώ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω εν συντομία. Προφανώ οι αναφορέ αυτές θα μείνουν ανοιχτέ, και θα στείλουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όλες αυτές τις συστάσεις της διερευνητικής μας αποστολής το ίδιο θα γίνει και προ την αρμόδια εισαγγελία και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση και θα περιμένουμε να δούμε έπειτα πώ θα εγκριθεί και πότε θα εγκριθεί το νέο αυτό νομοσχέδιο από το Ισπανικό Κογκρέσο. Το Μάιο του 2019 μα είπαν θα γίνει αυτό. Αυτή η πληροφορία που έχουμε επί του παρόντο. Θα ζητήσουμε μια επίγουσα, επίγουσα εφαρμογή τη νομοθεσία αυτή. Λοιπόν, επί του παρόντος νομίζω ότι αυτά μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως την Καθολική Εκκλησία για παράδειγμα, να ανταποκριθούν πραγματικά στις προσδοκίες των πολιτών, προκειμένου να επέλθει και αυτή η ευκταία συμφιλίωση. Και αυτό ουσιαστικά ισχύει και για όλους μας. Όλοι θα πρέπει να καταφέρουμε να συνεισφέρουμε με τρόπο θετικό, προκειμένου να περατωθεί με τρόπο ιδιαίτερα θετικό όλη αυτή η πολύ μακρά διαδικασία που ουσιαστικά αντιστοιχεί σε πολύ βαθιά ανθρώπινη οδύνη. Μόνο και μόνο τον έχει κανείς γνώση, να γνωρίζει τι έχει συμβεί, αποτελεί μεγάλο βήμα συμφιλίωσης. Και όπως σας είπα, μόνο η αλήθεια μας απελευθερώνει και ελπίζουμε ότι και στην περίπτωση αυτή αυτό θα συμβεί. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που ταξιδέψατε μέχρι τις Βρυξέλλες για μία ακόμη φορά. Να ευχαριστήσω πάλι βέβαια και την Τζουτ και όλους τους άλλους συναδέλφους, αλλά και τη Γραμματεία και ιδιαίτερα την Καρολίνα, η οποία εργάστηκε πολύ σκληρά για τις υποθέσεις αυτές. Και σας καλώ τώρα να περάσουμε στην επόμενη αναφορά, αλλά σας αφήνω λίγο χρόνο ώστε να καταφέρετε να αποχωρήσετε και να πάμε και εμείς στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. is Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, ας πάρουμε βαθιά ανάσα και ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη το υπαριθμό 31, αναφορά 0154 κάθετο 2018, όσον αφορά την επιτσίμαση των τροφίμων και τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, ευρωπαϊκό κανονισμό για τι ετικέτε που δείχνουν την προέλευση των τροφίμων. Βλέπετε ότι η Επιτροπή μα ασχολείται με τεράστια γκάμα θεμάτων. Περνάμε στην εντελώ διαφορετικό θέμα τώρα με αυτή την αναφορά. Θα ήθελα να καλωσορίσω καταρχά τον αναφέροντα, τον κύριο Ρομπέρτο Μονκάλβο, στον οποίο δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Καλημέρα σας. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αναφορών Κυρία Πρόεδρε Βίκστρομ, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλημέρα σας. Πραγματικά όντως πρέπει να πάρουμε βαθιά ανάσα για να αλλάξουμε θέμα μετά τις ιστορίες, τις τραγικές, τις οποίες ακούσαμε πριν από λίγο. Πρέπει όμως να το κάνουμε, να προσπαθήσουμε και να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, για τα τρόφιμα, για την προέλευση των τροφίμων, την επισήμανση των τροφίμων και για την καμπάνια Stop Chibo Falso, σταματήστε τα τις ψευδείς πληροφορίες για τα τρόφιμα, μια εκστρατεία την οποία ξεκίνησε η Συνομοσπονδία Ιταλικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Παραγωγής Τροφίμων που έχει συλλέξει πάρα πολλές υπογραφές. Πέρυσι τον Ιανουάριο ξεκινήσαμε τις εργασίες για την αφορά αυτή όταν γινόταν τότε και η δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού σε σχέση με τον κανονισμό 1169 του 2011. Αυτό το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού ήδη από τότε δεν μας έβρισκε σύμφωνους. Θεωρούσαμε ότι απήχε πάρα πολύ από τις απαιτήσει τόσο των γεωργών όσο και των Εβραίων πολιτών. Απαιτήσει τι οποίε έχει τονίσει πάρα πολλέ φορέ και έχει υποστηρίξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίω αυτή η θητεία του Κοινοβουλίου, όσον αφορά την υποχρεωτική επισήμανση τη πρόέλευση των τροφίμων, των γεωργικών τροφίμων. Συνεπώ, ήδη εμεί από τότε, από την εποχή τη διαβούλευση, αρχίσαμε την συλλογή υπογραφών για την αφορά αυτή. Σταματήστε τις ψευδείς πληροφορίε για τα τρόφιμα. Παράλληλα, με το σχέδιο αυτοεκλογιστικού κανονισμού, προχώρησε η δικασία αυτή και τελικά καταλήξαμε στον εκτελεστικό κανονισμό 775 του 2018, ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει από το 2020 και μετά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στη δική μας την αναφορά, ούτε τελικά στις απαιτήσει που αυτή εμπεριείχε όσον αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες και τους Ευρωπαίους γεωργούς. Και επίσης ο κανονισμός αυτός δεν ανταποκρίνεται καν στις απαιτήσει των ίδιων των κυβερνήσεων, των ίδιων των κρατών μελών, που αποφάσισαν, ιδίω για την επισήμανση των τροφίμων, να προτιμήσουν κυρίω την εθνική νομοθεσία. Υπάρχουν ήδη 9 χώρε με τις τελευταίες ε, που ε, υπέβαλαν εθνικές προτάσεις όπως η Ισπανία και η Αυστρία. Χώρες οι οποίες θέλουν να έχουν τελικά την δική τους εθνική νομοθεσία όσον αφορά την επισήμανση των τροφίμων. Εμείς αυτό το οποίο λέμε με την αναφορά είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε πραγματικά ένα ποιοτικό άλμα όσον αφορά την επισήμανση των γεωργικών τροφίμων για όλα τα γεωργικά τρόφιμα και είναι σαφές για μας πλέον ότι χρειαζόμαστε σαφείς και εναρμονισμένους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να λοιπόν για ποιο λόγο τους τελευταίους αυτούς μήνες και ιδίω από το Σεπτέμβριο και μετά, θεωρήσαμε λοιπόν χρήσιμο το ζήτημα της επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά δηλαδή τον τόπο προέλευσης και τη χώρα προέλευσης ότι θα έπρεπε αυτό να λάβει μια ευρωπαϊκή πλέον διάσταση ως ζήτημα και να μην αποτελεί πλέον μόνο ένα ιταλικό ζήτημα. Γιατί εντάξει, το Stop Cibo Falso, η καμπάνια αυτή ξεκίνησε στην Ιταλία, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό να λάβει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Και γι' αυτό το λόγο θελήσαμε να περάσουμε το θέμα αυτό μέσω μια μιας ευρωπαϊκή πρωτοβουλία των πολιτών. Ήδη τον Οκτώβριο στη Ρώμη άρχισε η συλλογή υπογραφών και έχουμε μπροστά μας πλέον ένα χρόνο για να καταφέρουμε να επιλέξουμε τις απαραίτητες υπογραφές και συνεργαζόμαστε ήδη με πάρα πολλούς άλλους ομόλογους φορείς σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το οποίο ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να κάνει αυτό το οποίο δεν έκανε με τον κανονισμό 1169 του 2011, τουλάχιστον να το κάνει τώρα μέσω του εκτελεστικού κανονισμού 775-2018, να έχουμε δηλαδή ένα σύστημα το οποίο να προβλέπει πλέον ένα υποχρεωτικό σύστημα, γιατί το σύστημα είναι θελοντικό αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα ολοκληρώνοντα το σημείο αυτό να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας και όλους τους Ευρω... ευρωβουλευτές που υποστήριξαν την Ιταλική μας καμπάνια, τον Αλμπέρτο Τσίριο, όλους ιδιαίτερα που μας πλαισίωσε πολύ επικοδομητικά σε όλη αυτή την πορεία μας, την Ελονόρα Εύη επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω, δύο ευρωβουλευτέ οι οποίοι αποφάσισαν να επαναφέρουν την αφορά αυτή στην Επιτροπή μόλον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είχε πει ότι προτίθεται να κλείσει την ανάλυση που κάνει για αυτέ τι αναφορέ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι συζητάμε δύο ζητήματα την υποχρεωτική επισήμαση της πρόλευσης των τροφίμων, όλων των τροφίμων και συζητάμε παράλληλα και τον εκτελεστικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στην υποχρεωτική αναφορά της προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού του τροφίμου όταν η προέλευση του, του πρωταρχικού συστατικού είναι διαφορετική από την προέλευση του συνολικού τροφίμου. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, το οποίο έθεσε ο αναφέρον, πρέπει να σας πω ότι η υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα κατά τη διάρκεια του κανονισμού για τις πληροφορίες που θα πρέπει να φέρουν τα τρόφιμα. Είχε διχάσει τότε αυτό τα κράτη-μέλη. Πολλά κράτη-μέλη ήταν υπέρ τη χρησιμοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια υποχρεωτική επισήμανση πρόλευση όλων των τροφίμων ή για κάποια προϊόντα, ενώ άλλα κράτη-μέλη πάλι ήταν κατά της πρότασης αυτής για λόγους που είχαν να κάνουν με το κόστος του εγχειρήματο αυτού ή λόγω ζητημάτων που είχαν να κάνουν με την εσωτερική αγορά. Το αποτέλεσμα λοιπόν διαπραγματεύσεων αυτών ήταν ότι αποφασίσαμε εμείς να διευρύνουμε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της επισήμανσης των τροφίμων για κάποια προϊόντα και ιδίω για το κρέος, τον οπό κρέας, ενώ για κάποια άλλα προϊόντα αποφασίσαμε να υποβάλουμε εκθέσεις και να βλέπουμε κάθε φορά κατά περίπτωση αν πρέπει να επεκτείνουμε την υποχρέωση αυτή και σε άλλους τομείς όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα μη μεταποιημένα προϊόντα και το καθεξής έκανε όλη αυτή την εργασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέβαλε όλε αυτέ τι εκθέσει και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η εθελοντική τελικά προσέγγιση ήταν πολύ καλύτερη από την υποχρεωτική προσέγγιση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε και με την εφαρμογή κάποιων άλλων απαιτήσεων που είχαν ω στόχο να πλαισιώσουν τις εθελούσιες επισημάνσεις προέλευσης τροφίμων έτσι ώστε ο καταναλωτής να ενημερώνεται όταν η χώρα ή ο τόπος προέλευσης που αναφέρεται για ένα τρόφιμο διαφέρει από εκείνο του πρωταρχικού συστατικού του τροφίμου αυτού. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει λοιπόν μια κάποια ευελιξία και ακούσαμε ότι αναφέροντες έχουν παραπονεθεί για το ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο επίπεδο λεπτομέρεια. Παρ' όλα αυτά, όμω, μόνο και μόνο η αρχική νομοθετική πράξη προβλέπει την απαραίτητη αυτή ευελιξία, προκειμένου οι αρμόδιοι φορεί παραγωγή να αναφέρουν τον τόπο προέλευση του πρωταρχικού συστατικού με τρόπο συγκεκριμένο ή να λένε απλώ ότι η χώρα ή ο τόπο προέλευση που αναφέρεται για ένα τρόφιμο διαφέρει από εκείνο του πρωταρχικού του συστατικού. Επίση, ε, οι αναφέροντε ε, μας είπαν ότι δεν υπάρχουν ε, οι απαραίτητοι κανόνες που να καλύπτουν ακόμα και τα κατοχυρημένα εμπορικά σήματα ή τα προϊόντα που φέρουν προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να πω ότι ο εκτελεστικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν εξαιρεί, δεν αποκλεί, όπως είπε ο αναφέρον, τα εμπορικά σήματα ή τις γεωγραφικές ενδείξεις, απλώς αναβάλει, μεταθέτει την εφαρμογή των κανόνων αυτών για τις κατηγορίες αυτές και αυτό γίνεται για τους λόγους που εξηγούμε στις ιδεολογικές σκέψεις, συγκεκριμένα την 6 και την 7. Λέγεται εκεί στι ιδεολογικές αυτές σκέψεις του κανονισμού ότι και τα εμπορικά σήματα και οι γεωγραφικέ ενδείξει εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού τώρα. Η μελέτη αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάλυψε συγκεκριμένα τα εμπορικά σήματα ή τι γεωγραφικέ ενδείξει και γι' αυτό ακριβώ το λόγο αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσωρινά να εξαιρεθούν οι δύο αυτέ κατηγορίε μέχρι να καταλήξουμε σε συγκεκριμένου κανόνε οι οποίοι θα υιοθετηθούν κάποια στιγμή στο μέλλον. Συνεπώς, θεωρούμε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ως έχει είναι απολύτω ικανοποιητικό και όντως μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου ενδεχομένω ένα καταναλωτή να πέσει θύμα παραπλανητικών πληροφοριών όσον αφορά τον τόπο προέλευση τροφίμων. Ξέρουμε ότι σε εθνικό επίπεδο ισχύουν κάποια εθελοντικά προσωρινά εθνικά συστήματα επισήμανση των τροφίμων, τα οποία αυτόματα όμως θα καταργηθούν περίπου το Μάιο του 2020, όταν θα αρχίσει υποχρεωτικά για όλα τα κράτη-μέλη να ισχύει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, το πεδίο εφαρμογή αυτών των εθνικών κανόνων είναι πολύ πιο ευρύ από το πεδίο εφαρμογή που προβλέπει ο δικό μα εκτελεστικό κανονισμό. Καλύπτει ουσιαστικά όλε τι περιπτώσει εκείνε όπου σε εθνικό επίπεδο πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται ο τόπο προέλευση, ιδίω για το κρέα και για τα γαλακτοκομικά. Δεν αναφέρεται δηλαδή η εθνική νομοθεσία ή οι εθνικέ νομοθεσίε μόνο στην περίπτωση εκείνη όπου ο τόπο προέλευση που αναφέρεται για ένα τρόφιμο διαφέρει από εκείνο του πρωταρχικού του συστατικού. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι στην αίθουσα, αλλά φαντάζομαι όλο και κάποιο Ιταλό θα ήθελε το λόγο. Ελεονόρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για την αναφορά αυτή, η οποία αγγίζει ένα θέμα το οποίο αφορά όλους εμάς τους Ευρωπαίους πολίτες. Τα τρόφιμα, τα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε λοιπόν δυστυχώς δεν φέρουν όλες τις ακριβείς πληροφορίες που θα έπρεπε να αναγράφονται πάνω στις συσκευασίε. Και αυτό το λέω ξεκάθαρα. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες, η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν μας επιτρέπει να μπορούμε να κάνουμε μία σίγουρη, τεκμηριωμένη, συνειδητή επιλογή όσον αφορά τα τρόφιμα, έχοντας την πεποίθηση ότι τα τρόφιμα αυτά είναι ασφαλή πολύ συχνά τα όσα αναγράφονται στις επισημάνσεις των τροφίμων δεν είναι σαφή, είναι αρκετά ελλειπή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει τόσο πολύ στον εθελοντικό αυτό χαρακτήρα τη επισήμανση των τροφίμων. Και έρχεται μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μα λέει ότι αυτό είναι και βέλτιστη πρακτική, την οποία θα πρέπει να υιοθετήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Μα δεν ισχύει αυτό. Και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, αλλά και το 70% των ε, Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι συμμετείχαν μάλιστα σε μία έρευνα του ε, Ευρωβαρομέτρου. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών λέει ότι θέλει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη χνηλασιμότητα όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία αγοράζουν κυρίω τα τρόφιμα. Και προκαλεί εντύπωση κιόλα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελαφριά την Καρδία έρχεται και μας μιλάει εδώ πέρα για τον εκτελεστικό κανονισμό που εγκρίθηκε φέτος λέγοντάς μας ότι αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου και ότι ξαφνικά αυτή τη στιγμή δημιουργείται και υποχρέωση για την αναφορά της προέλευσης του ποταρχικού συστατικού. και παράλληλα δημιουργεί πάρα πολλές εξαιρέσεις που αφορούν τα εμπορικά σήματα, που αφαιρούν τις γεωγραφικές ενδείξεις και δικαιολογεί τι εξαιρέσει επίση αυτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγοντά μα ότι μην ανησυχείτε, τι τομεί αυτού θα του καλύψουμε κάποια στιγμή και στο μέλλον, όταν γίνουν οι απαραίτητε αναλύσει και απαραίτητε έρευνε. Τίποτα δεν μα λέει ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ θα εξελιχθεί πραγματικά ο ενισχύει κανονισμό. Και συμφωνώ απόλυτα με τι ανησυχίε που εγείρουν οι αναφέροντε, όχι μόνο για τον κανονισμό, αλλά και για το σχέδιο του εκτελεστικού κανονισμού. Πρόβλημα έχει και ο αρχικός ο κανονισμός, ο 1169 του 2011, ο οποίος είναι πολύ ελλειπής, πολύ ασθενή σε κανονισμό και σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάζει διασφαλίσει για τα χένια τα οποία θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Καλύτερη εχνηλασιμότητα, περισσότερε γνώσει όσον αφορά την προέλευση των τροφίμων. Επίσης, είδαμε με πόσο μεγάλη καθυστέρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να σκουμποθεί και να κάνει κάτι Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να κινητοποιηθεί όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο το έχει κάνει πάρα πολλέ φορέ κατά τη διάρκεια τη θητεία αυτή, με αμέτρητα ψηφίσματα τα οποία έχουμε υποβάλει, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο συγκεκριμένε πληροφορίε, αλλά και μέσω των ίδιων των πολιτών. Οι ίδιοι Ευρωπαίοι πολίτε, όπω βλέπετε, χρησιμοποιούν τόσα πολλά μέσα κοινωνική συμμετοχή σε σύμπραξη, προκειμένου πραγματικά να καταφέρουν και αυτοί να προωθήσουν περισσότερο το ζήτημα αυτό. Είναι επίση ε, πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώ θα εξελιχθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που ήδη έχει ξεκινήσει φέτο. Εγώ θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τον εκατομμύριο υπογραφέ και να αποχρεώσουμε έτσι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σημειώσει απτά βήματα προόδου. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να πω ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, σε ένα σημείο καμπής. Δεν έχει την πολυτέλεια να μην ακούει πλέον τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν έχει την πολυτέλεια να παραβλέπει συνειδητά τι πραγματικέ ανησυχίε των πολιτών. Γιατί αυτό που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή είναι η ίδια εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολίτε οι οποίοι απαιτούν όχι μόνο να προστατευτεί η υγεία του, αλλά απαιτούν μεγαλύτερη ποιότητα και περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα τα οποία αγοράζουν και προφανώς και για τα τρόφιμα. Πραγματικά λυπάμαι που δεν έχουμε και ευρωβουλευτές από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ο αγώνας αυτός που δίνουμε δεν είναι μόνο ιταλικός, είναι και ευρωπαϊκός αγώνας. Ένας αγώνας προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει κανόνες οι οποίοι πραγματικά ανατάσσονται υπέρ των πολιτών. Θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Ελεονόρα. Ο κύριος Τσίριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ ευαίσθητο και λεπτό το θέμα, γιατί ουσιαστικά υπερβαίνει τον τομέα των τροφίμων έχουμε μία από τις περιπτώσεις εκείνες όπου φαίνεται πλέον ξεκάθαρα πώς καταφέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χάσει την αξιοπιστία της απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί υποπέπτει η ίδια, υπο, υποπίπτει η ίδια σε αντιφάσεις. Λέμε ότι θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρεσβεύει παντού ότι θέλει περισσότερη διαφάνεια. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέμε ότι θέλουμε να είμαστε ένα οίκο διαφάνεια. Επιγραμμικά διαβιβάζουμε τα εγγραφά μας, μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου οι συζητήσεις μας οι Ευρωπαίοι πολίτε το μόνο το οποίο θέλουν αυτή τη στιγμή είναι να γνωρίζουν τι τρώνε. Και για αυτό το ουσιαστικότατο και βασικό θέμα έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι κοιτάξτε το σύστημα το οποίο σας προτείνει είναι θελοντικό. Δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται παντού ο τόπο προέλευση των τροφίμων. Μα πώ μπορούμε να αντιδρούμε έτσι για ένα ζήτημα το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Εγώ θέλω να ξέρω τι τρώω, είμαι αυτό που τρώω. Ως Ευρωπαίοι πολίτες αυτό το οποίο ζητάμε είναι να έχουμε τι απαραίτητες πληροφορίε, να είμαστε ενήμεροι για το τι καταναλώνουμε. Θέλουμε η Ευρώπη, η οποία πρεσβεύει τόσο πολύ τη θεωρία αυτή τη διαφάνεια, να είναι πραγματικά διαφανή και σε σχέση με τι πληροφορίε που παρέχει στου πολίτε για τα τρόφιμα, για τα αγροτικά προϊόντα τα οποία οι πολίτε καταναλώνουν. Το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο δεν έχει εγκρίνει του κανόνε αυτού, αλλά ότι φαίνεται τελικά να μην αφογκράζεται καν τις ανάγκες των πολιτών, αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Έχουμε τον κανονισμό και έχουμε έπειτα και τον εκτελεστικό κανονισμό που τίθεται ότι μας δίνει και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Και απευθύνομαι τώρα και ως εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο άνθρωπος ο οποίος παράγει ένα τρόφιμο, ένα προϊόν, το οποίο φτάνει σε μία χώρα, ε, θα πρέπει όχι αναγκαστικά ο αυτός ο ίδιος να προστατεύεται, αλλά να δούμε πώς θα καταφέρουμε να, θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες που καταναλώνουν το προϊόν αυτό. Αρκεί να βάλει κανείς την Ιταλική σημαία πάνω στη συσκευασία ενός οποιοδήποτε προϊόντος για να παραπλανήσει τελικά τους καταναλωτές, οι οποίοι νομίζουν ότι καταναλώνουν Ιταλικό προϊόν, πράγμα το οποίο δεν ισχύει στην πράξη. Και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Αν επισήμως δεν αναγράφεται η προέλευση του συγκεκριμένου προϊόντος δεν προστατεύουμε τον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίο δεν γνωρίζει τελικά τι τρώει, αλλά δεν προστατεύουμε και τους μικρούς παραγωγούς, τις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν πραγματικά τοπικά προϊόντα και οι οποίες θα θέλανε να αναγράφεται όντως η προέλευση, η αυθεντική προέλευση του προϊόντος. Νομίζω λοιπόν ότι ή θα πρέπει ο κανόνα να ισχύει υποχρεωτικά για όλου, ακόμα και τα προϊόντα τα οποία μα έρχονται από την Αμερική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική, να αναγράφεται υποχρεωτικά η προέλευση των τροφίμων. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα είμαστε ποτέ ανταγωνιστικοί. Γιατί αν νομίζουμε ότι μπορούμε στο γεωργικό τομέα να συναγωνιστούμε τι τεράστιε ποσότητε που παράγουν τρίτες χώρε, έχουμε χάσει εξ αρχή το παιχνίδι. Εμεί μπορούμε να επενδύσουμε μόνο στην ποιότητα. Αυτό αν θέλετε είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Η ποιότητα όμως έχει να κάνει και με την επισήμανση των τροφίμων, δηλαδή με το τι αναγράφεται όσον αφορά την χώρα ή τον τόπο προέλευσης ενός τροφίμου. Και πραγματικά μου είναι ασύλληπτο το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το συνειδητοποιεί το πράγμα αυτό. Αν τώρα υπάρχει ένα μικρό κόστος προκειμένου μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με την υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων, ε, τότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου να βοηθήσει τους μικρούς παραγωγούς για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες. Δεν μπορεί αυτό να αποτελεί από μόνο το εμπόδιο. Διότι, όπως σας είπα, Πρέπει να προστατεύσουμε τα προϊόντα μας, όχι μόνο τα ιταλικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο παραποίηση, όπως ξέρετε, σε πάρα πολλέ χώρες. Αυτό ισχύει και για τα ισπανικά, τα γαλλικά προϊόντα και για τα προϊόντα πολλών άλλων χωρών τη Ένωση. Ευχαριστώ. Η διαφάνεια είναι αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε ακριβώ, όπω λέτε και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ε, δεν γίνεται κάποιο στην Ιταλία να παίρνει, ε, να αγοράζει λάδι από την Ισπανία και να βάζει πάνω απλά μια ετικέτα που γράφει Ιταλικό λάδι. Θα πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχεται και επίσης ε, ε, Ιταλικά προϊόντα τα οποία γίνονται, κατασκευάζονται στην Κίνα και τα φέρνουν στη συνέχεια στην Ιταλία και πολλούνται με την ετικέτα Made in Italy. Ε, ο κύριος Ταμπονάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί με κάλυψαν οι συναδελφοί μου οι οποίοι πραγματικά αναφέρθηκαν με κάθε δυνατή λεπτομέρεια σε όλες τις πτυχές του ζητήματος. Μιλήσαμε για την προστασία της εσωτερική αγοράς. Η εσωτερική αγορά είναι μια αγορά ελεύθερων συναλλαγών. θα πρέπει εδώ πέρα πραγματικά να δούμε πώς επηρεάζουμε την ελεύθερη επιλογή του καταναλωτή, του Ευρωπαίου πολίτη. Ο πολίτης θα πρέπει να είναι ελεύθερος να μπορεί να επιλέγει τα προϊόντα εκείνα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. Και αυτό συνδέεται με την αρχή της διαφάνειας. Ελευθερία και διαφάνεια είναι δύο αλληλένδετες για μένα έννοιες πραγματικά θα πρέπει να καθοδηγούν πάντα τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφώς θα πρέπει να εργαστούμε για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης περνά σίγουρα μέσα από τα τρόφιμα. Διότι τα τρόφιμα αντιστοιχούν και στην υγεία, τη δημόσια υγεία. Το να γνωρίζουμε από πού προέρχεται ένα προϊόν, αν προέρχεται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ή από συγκεκριμένο κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αυτό θα πρέπει να εγγράφεται σε συγκεκριμένους κανονισμούς. Κανονισμούς οι οποίοι επίσης να υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να αναγράφουν και τυχόν ζυζανιοκτώνα ή άλλα χημικά προϊόντα τα οποία να περιέχονται στην, στα προϊόντα αυτά. Επομένως μιλάμε αυτή τη στιγμή για ελευθερία επιλογής, μιλάμε για διαφάνεια αλλά και προώθηση περισσότερο των κρατών εκείνων τα οποία κάνουν τις πιο ποιοτικέ επιλογές. Να υπάρχει απαραίτητη αξιοκρατία. Υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας όμως, οι κλιματικές αλλαγές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται μια αναγραφή του τόπου προέλευσης προκειμένου ο Ευρωπαίος πολίτη να μπορεί να επιλέγει το προϊόν εκείνο το οποίο συμβάλλει στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ακριβώς επειδή είναι το προϊόν εκείνο το οποίο παράγεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του και δεν είναι ένα προϊόν το οποίο έχει εισαχθεί από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ένα προϊόν δηλαδή με ένα οικολογικό, αν θέλετε, περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα προϊόν το οποίο έχει οδηγήσει σε μειωμένε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί όχι μόνο οι Ιταλοί αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν ζητήσει την αγραφή όλων αυτών των ενδείξεων. Ευχαριστώ πολύ. Να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Μονκάλβο, τον αναφέροντα. Σας ευχαριστώ και να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές που πήραν το λόγο. Να ευχαριστήσω επίσης την Πρόεδρο για τα όσα είπε. Πιστεύω πραγματικά ότι ακόμα και αυτά που μας είπε σήμερα το πρωί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύει το ότι δεν θέλει τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες όχι μόνο των Ιταλών αλλά γενικότερα των Ευρωπαίων πολιτών. Σας πενθυμίζω ότι ο κανονισμός 775 του 2018 θα αρχίσει να ισχύει με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με αυτά τα οποία αναγράφονται στον κανονισμό 1169 του 2011. Με καθυστέρηση λοιπόν έρχεται ο εκτελεστικός κανονισμός και δεν μα ικανοποιεί το περιεχόμενό του. Επομένως είμαι πεπισμένο για αυτό που σα είπα πριν από λίγο. Αυτές οι 120.000 υπογραφέ της καμπάνιας Stop Cibo Falsi στην Ιταλία αποτελούν μόνο την αρχή της προσπάθειας για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία των πολιτών προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να έχουμε αυτό το 1 εκατομμύριο υπογραφέ που απαιτούνται από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προκειμένου να υποχρεωθεί πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έστω η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τροποποιήσει ακόμα και το βασικό κανονισμό, των 1169, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια νομοθεσία που θα ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων που προέρχονται, τροφίμων και όλων των γεωργικών προϊόντων ουσιαστικά. Ελπίζω ότι ε, θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ολοκλήρωση της συλλογή των υπογραφών αυτών προτού αρχίσει να ισχύει ο εκτελεστικός κανονισμός 775-2018. Να ευχαριστήσω πραγματικά την Επιτροπή Αναφορών για όλο τον χρόνο που μας αφιέρωσε σήμερα και ελπίζω ειλικρινά ότι το πολιτικό αυτό θέμα της επισήμανσης των τροφίμων θα εξακολουθεί να απασχολεί και να αξιολογείται εδώ πέρα από τους βουλευτές Επιτροπής Αναφορών τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ολοκληρώσουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή και να την ε, προωθήσουμε στη συνέχεια στην Envy και την Άγκρη για να γνωμοδοτήσουν. Από την Envy έχουμε ζητήσει ήδη γνωμοδότηση, δεν έχουν ποτίσει ακόμα, οπότε θα στείλουμε μια υπενθύμηση ότι ανυπομονούμε να λάβουμε την γνωμοδότησή τους και στην Άγκρη όμως θα πρέπει να το στείλουμε το θέμα για να δούμε τι θα μας απαντήσουν και ίσως ε, θα μπορούσαν να παρουσιάσουν ε, έναν τρόπο για να προχωρήσουμε. Ελεονόρα. Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι ακόμα. Ένα μικρό σχόλιο, κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε επίσης ε, τον ασταλή αναφορά αυτή και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και μια πρόταση για το μέλλον. Θα μπορούσαμε ε, να κανονίσουμε μια δημόσια ακρόαση ως ε, κληροδότημα αυτών των αναφορών ε, για ε, την ε, επόμενη θητεία. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να λάβουμε δεσμευτικές αποφάσεις για την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι μια πρόταση, ένα πολιτικό μήνυμα, το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό να πάρουμε την κληρονομιά αυτή της αναφοράς και να μεταφερθεί και στο επόμενο Κοινοβούλιο. Ναι, φυσικά μπορούμε να το στείλουμε και στην ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Έτσι θα το κάνουμε λοιπόν. Τώρα όσον αφορά την οργάνωση, γνωρίζετε ότι ο πολιτική σας ομάδα μπορεί να το κάνει μέσω συντονιστών. Εκεί λαμβάνουμε τις ε, αποφάσεις ε, σε, για ζητήματα σχετικά με ακροάσεις Εφόσον είστε η συντονίστρια λοιπόν της ομάδας σας μπορείτε να παρουσιάσετε την ιδέα αυτή και να δείτε αν βρίσκει αότα. Είμαι ακριβέστατη, 12 και 30 θα τελειώναμε για σήμερα. Σας εύχομαι όλους λοιπόν καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα καλό μεσημεριανό γεύμα.